Ladies Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ, θα ξεκινήσουμε αμέσω. Καλημέρα και καλωσορίσατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας. Η ημερήσια διάταξη διανεμήθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Θα ήθελα να σε επενθυμίσω ότι μεταδίδεται από το διαδίκτυο η συνεδρίαση και υπάρχει διερμηνία στις γλώσσες ε, των μελών της Υποπιτροπής Ασφάλειας και Άμυνας. Παρακαλώ να εγκριθεί η μερίσια διάταξη. Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνεται συνεπώς η μερίσια διάταξη. Υπάρχει χρόνος μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, αρκετός χρόνος, στις 12.30 θα τελειώσουμε. Υπάρχει συνεπώς χρόνος για να διατυπώσετε τυχόν επιφυλάξεις όσον αφορά ε, την συνεδρίαση της 26 Φεβρουαρίου. Εάν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις, τότε θα θεωρηθούν τα πρακτικά ότι έχουν εγκριθεί. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω και τους προσκεκλημένους μας, ε, τον προδευτή Γιάτσεφ Μπιλίτσα, κύριο σύμβουλο και ειδικό απεσταλμένο για τη μη διάδοση και τον αφοπλισμό ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και του δίνω αμέσως το λόγο για να με συνημερώσει σχετικά με την θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την συντονισμένη θέση μας. Δεδομένου ότι τα κράτη-μέλη έχουν ε, προσυπογράψει την ε, συνθήκη για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων και θα μας μιλήσει για την αναθεώρηση της ε, διάσκεψης επί ε, της συνθήκης των ε, διάδοσης εμπειρικών όπλων που έλαβε χώρα φέτος, στην αρχή του έτους. Παρακαλώ Κύριε Μπρίτσα, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε για την ανταλλαγή απόψεων όσον αφορά την αναθεώρηση ε, τη συνθήκη μη διάδοση που πρόκειται να λάβει η χώρα στην έδρα των ΗΕ στη Νέα Υόρκη μεταξύ 27 Απριλίου και 22 Μαου 2015. αυτή η διάσκεψη αναθεώρησης είναι χωρίς αμφιβολία η πιο σημαντική εκδήλωση ε, στο ημερολόγιο, στην ατζέντα ε, της ε, μη διάδοσης των πυρηνικών όπλων και του φοπλισμού. Και αυτό έρχεται μετά από μια συζήτηση που έγινε στις 10 Φεβρουαρίου του 2015 στο Στρασβούργο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου η κυρία Φεντρίκα Μογκαρίνη είχε συμμετάσχει επίσης. Ε, έγινε αντικείμενο ακρόασης ε, στην ΣΕΝΤΕ τον Ιανουάριο, στις 29 Ιανουαρίου, με τη συμμετοχή του συναδέλφου μου, του επικεφαλής ε, της, του τμήματος και την κυρία Κλάρα Γκάνσλατ. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτή τη διάσκεψη προετοιμάζεται τώρα ε, στα πλαίσια της ΕΕΔ και μεταξύ των κρατών μελών. Προγραμματίζεται να ε, υπάρξει συνημερίσια διάταξη ε, του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων του Απριλίου 2015. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω τι εξή παρατηρήσει, χωρί να προδικάσω τα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Η προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στον αποκλεισμό ε, και στη μη διασπορά ε, των ε, όπλων μαζική καταστροφή καθοδηγείται από την αρχή του αποτελεσματικού πολυμερισμού που περιλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταβάλει κάθε προσπάθεια να εξασφαλίσει αφενό την παγκοσμιοποίηση και αφετέρου την αποτελεσματική υλοποίηση ε, των αντιστοίχων διεθνών συνθήκων και άλλων νομικών οργάνων συμπεριλαμβανομένης της μια διασπόρά. Επίση, υποστηρίζουμε οικονομικώς τι διεθνείς οργανώσει, επιφορτισμένες με την εφαρμογή τους όπως ε, τον Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας IEA. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη όσον αφορά ε, την διασπορά των πυρηνικών όπλων που είναι ακρογωνιαίο λήθος όσον αφορά ε, τον πυρηνικό φοπισμό σύμφωνα με το άρθρο 6 της συνθήκης που είναι αποτελεσματικό στοιχείο για την ανάπτυξη των, ε, της εφαρμογής πυρηνικής ενέργειας για πυρηνικούς σκοπούς. Γι' αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να αποτελέσει αυτή τη συνθήκη μια βασική προτεραιότητα για την ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας και σταθερότητας. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να επαναλάβουμε ε, την υποστήριξη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τρεις πυλώνες της συνθήκης και για την εφαρμογή όλων των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί ε, στις προηγούμενες διασκέψεις αναθεώρησης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να προωθεί μία ολοκληρωμένη, ισορροπημένη και ουσιαστική πλήρη εφαρμογή ε, του σχεδίου δράσης 2010 που περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για τον αφοπλισμό, τον πυρηνικό αφοπλισμό, τη μη διασπορά και τις, τις ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας. Εξασφαλίζοντας ε, την εφαρμογή των 64 δράσεων του σχεδίου δράσης είναι μια συλλογική ευθύνη όλων των κρατών μερών που έχουν συνυπογράψει τη συνθήκη. Χωρίς αυτό τον κύκλο να θεώρηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση μαζί με ε, τα κράτη-μέλη υποστηρίζουν την εφαρμογή της συνθήκης όχι μόνο με διπλωματικά μέσα, αλλά με κατάρτιση ε, και βοήθεια και συνεπώς συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της συνθήκης. Όσον αφορά ε, τον πυρηνικό αφοπλισμό, με την δέσμευση των κρατών μέλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με το άρθρο 6 της συνθήκης και υπογραμμίζουμε την ανάγκη συγκεκριμένη πρόοδου στον τομέα, κυρίως ε, μια γενική μείωση ε, των αποθεμάτων πυρηνικών όπλων. Μέχρι τώρα έχουν γίνει μειώσεις λαμβάνοντας υπόψη την ειδική ευθύνη των κρατών μελών που κατέχουν τα μεγαλύτερα οπλοστάσια, δηλαδή την Ρωσική Ομοσπονδία, τις ΗΠΑ. Ε, σε αυτά τα πλαίσια καλωσορίζουν επίσης τις ενδείξεις πρόοδου στην εφαρμογή της νέας συνθήκης START και παροτρύνει τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν σε μεγαλύτερες μειώσεις του πυρηνικού ε, οπλοστασίου τους, συμπεριλαμβανομένων στρατηγικών, μη στρατηγικών, αναπτυγμένων και μη αναπτυγμένων όπλων καλωσορίζει και παροτρύνει ε, την σύγκληση της, ε, των διασκέψεων P5 καθώς και τις ε, δραστηριότητες επαλήθευσης και ελέγχου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται στον αφοπλισμό και τον έλεγχο των εξοπλισμών και για αυτό το λόγο υπογραμμίζει την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες όσον αφορά τον αφοπλισμό. δεδομένου ότι δεν έχει προχωρήσει αυτός ο τομέας, αυτό προβληματίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να, να επαναλάβουμε ότι αυτή η διάσκεψη είναι ε, πολύ σημαντική ε, και ε, γι' αυτό παροτρύνουμε στην ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων για τον αφοπλισμό και για τη συνθήκη που απαγορεύει την παραγωγή σχάσιμων υλικών. εξακολουθούμε να προωθούμε αυτό το στόχο μέσω διπλωματικών διάβλων. Σημειώνουμε τις σοβαρές συνέπειες που έχουν σχέση με τη χρήση των πυρηνικών όπλων και υπογραμμίζουμε ότι όλα τα κράτη-μέλη έχουν ευθύνη να αποτρέψουν αυτά τα συμβάντα στα πλαίσια των συζητήσεων που γίνονται για τις συνέπειες ε, των πυρηνικών όπλων, διάφορες απόψεις διατυπώνονται, όπως στη διάσκεψη της Βιέννης για τις ε, ανθρωπικές επιπτώσεις των πυρηνικών όπλων που οργανώθηκε το Δεκέμβριο 2014 από την Αυστρία. Παρόλο ότι όλα τα κράτη-μέλη δεν είχαν λάβει μέρος σε αυτή την εκδήλωση, η πλειοψηφία των κρατών μελών που ήσαν παρόντα συμφώνησαν ότι μια σταδιακή προσέγγιση ήταν ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί ο πυρηνικός αφοπλισμός. Επ' αυτού πρότειναν πολλά ε, μονομερή, πολυμερή μέτρο και διμερή μέτρα, όπως ε, την ε, συνθήκη που απαγορεύει την παραγωγή σχασίμων υλικών για την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψη το περιβάλλον τη ασφάλεια, όταν γίνεται συζήτηση για τα πυρηνικά όπλα και τον πυρηνικό φοπλισμό. Για την μη διάδοση των πυρηνικών όπλων αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση τις μεγάλες προκλήσεις από τον τομέα που εξακολουθούν να συνιστούν απειλή στη διεθνή ασφάλεια και την ανάγκη να βρεθούν ειρηνικέ και διπλωματικές λύσεις. Υπογραμμίζουμε ότι η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να επαγρυπνεί και να είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει αυτέ τι προκλήσει και με αποφασιστικό τρόπο. Αναγνωρίζουμε ότι το σύστημα διασφάλιση είναι σημαντικό ε, στοιχείο ε, του καθεστώτο μη διάδοση πυρηνικών όπλων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει την μεγάλη ευθύνη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης. Για τα περιφερειακά θέματα πρέπει να υπογραμμίσουμε την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημιουργία μιας ζώνης απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη λύπη της επειδή μέχρι τώρα δεν μπόρεσε να συγκαλέσει μια διάσκεψη για τη δημιουργία μιας τέτοιας ζώνης ώστε να παρευρεθούν όλα τα κράτη της περιοχής. Υποστηρίζομαι τις προετοιμασίες που γίνονται και επίσης θα θέλαμε να συγχαρούμε αυτούς που την οργάνωσαν καθώς και τον φορέα διευκόλυνσης και την ομάδα του καθώς και τις άτυπες συναντήσεις που έγιναν ε, στην Ελβετία. Για να υποστηριχθεί αυτός ο στόχος, η Ευρωπαϊκή Ένωση οργάνωσε ε, πολλές εκδηλώσεις Track 2 ε, υπομορφή σεμιναρίων το 2011 και το 2012 στις Βρυξέλλες με αξιωματούχους των κρατών μελών της περιοχής. Επίσης οργάνωσε ένα σεμινάριο για τη δημιουργία ικανοτήτων όπου έγινε ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ εκείνων που διαπραγματεύονται τις απαλλαγμένες από πυρηνικά όπλα ζώνες. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να επαναβεβαιώσω τη σημασία που αποδίδει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην παγκοσμιοποίηση ε, της συνθήκης. Ζητήσαμε στα κράτη-μέλη που δεν το έχουν κάνει να προσχωρήσουν στη συνθήκη και αν να συμμορφωθούν στους όρους. Η... Στις 2 Απριλίου 2015 η ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος των ΗΕ και ο Υπουργός Εξωτερικών της, ε, του Ιράν έκαναν μια κοινή δήλωση στην Ελβετία και κατέληξαν σε λύσεις για να υπάρχει ένα κοινό πρόγραμμα δράσης για να εξασφαλίσουν ε, την πυρηνική χρήση του, ε, την ειρηνική χρήση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Οι εργασίες θα συνεχιστούν σε επίπεδο πολιτικό και μυρογνώμων για να συνταχθεί το κείμενο αυτού του κοινού ε, προγράμματος δράσης. Οι δύο πλευρέ έχουν δεσμευθεί να ολοκληρωθούν αυτέ οι προσπάθειε μέχρι τι 30 Ιουνίου. Είμαι βέβαιο ότι αυτή η σημαντική εξέλιξη θα έχει ε, σημαντική επίπτωση στην ατμόσφαιρα και στην έκβαση ε, τη διάσκεψης αναθεώρηση. Επίση στη Μέση Ανατολή η Ευρωπαϊκή Ένωση λυπάται επειδή η Συρία ακόμα δεν έχει συμμορφωθεί ε, με τη Συμφωνία των Ρητρών Διασφάλισης. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να υπογραμμίζει τις άλλες προκλήσεις που τίθενται όπως οι δοκιμές που γίνονται από, την δημοκρατική, από τη Δημοκρατία της Κορέας. Επίσης υπογραμμίζει τις ελληνικές χρήσεις της ενέργειας και η Ευρωπαϊκή Ένωση επαναβεβαιώνει ε, την ε, υποστήριξή της για τα αναφέρετα δικαιώματα όλων των χωρών να αναπτύξουν την πυρηνική ενέργεια για ειρηνικούς σκοπούς χωρίς διάκριση και σύμφωνα με τη συνθήκη. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσουμε στα κράτη-μέλη που έχουν υπογράψει συνθήκη, ώστε να αναπτύξουν με ευθύνη ε, τα πυρηνικά, ε, τις πυρηνικές χρήσεις, ε, τις πυρηνικές χρήσεις πυρηνικής ενέργειας. Η ενίσχυση της πυρηνικής ασφάλειας είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι σημαντικό στοιχείο της διευκόλυνσης της διεθνούς συνεργασίας. Η διάσκεψη κορυφής για την ασφάλεια έχει ως αντικείμενο να ενισχύσει την πυρηνική ασφάλεια, περιορίζοντα την απειλή της πυρηνική τρομοκρατία και εξασφαλίζοντα ότι όλα τα πυρηνικά ε, ε, ε, υλικά θα είναι ασφαλή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι δεσμευμένη σε αυτούς τους στόχου, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο της διάσκεψης και οι σημαντικέ ε, συνέπειε ε, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και παρατηρούμε όλα τα κράτη-μέλη να, ε, να συζητήσουμε με κοδηματικό τρόπο την αποτροπή των πυρηνικών ατυχημάτων. Και αν υπάρξουν ατυχήματα, τότε να μετριάζουν τα αποτελέσματα και η μόλυνση. Διακεκριμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Προφανώς πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτή η διάσκεψη θα λάβει χώρα με μία βάση ενός περιβάλλοντος δύσκολου για την ασφάλεια, όπου υπάρχουν μεγάλες απειλές και κίνδυνοι από το τρομακτικό σενάριο των τρομοκρατών που μπορεί να έχουν στα χέρια τους όπλα μαζικής καταστροφής μέχρι την επίθεση κατά της ασφάλειας, της εδαφικής ακαιρεότητας και της κυριαρχίας των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι πρόφαση για να μην ληφθούν μέτρα. Το αντίθετο μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Ένωση παροτρύνει όλες τις χώρες που έχουν προσυπογράψει τη συνθήκη να καταλήξουν σε επιτυχή έκβαση ώστε το αποτέλεσμα να είναι θετικό. Ο είπατε εκπρόσωπος έχει ε, επιβεβαιώσει ότι θα συμμετάσχει προσωπικά σε αυτή τη διάσκεψη, καθώς και αρκετοί Υπουργοί Εξωτερικών και ανώτεροι αξιωματούχοι από τα κράτη-μέλη μας. Προσωπικά ελπίζω ότι υπό την ικανή ηγεσία ε, του πρεσβευτή Κάος Φερούκη της Αλγερίας θα ολοκληρώσουμε αυτούς τους σημαντικούς στόχους. Μπορεί η Πρόεδρος να στηρίζεται στην υποστήριξή μας και μάλιστα πρόσφατα οργανώσαμε ένα σεμινάριο στην, στο Αλγέρι για την προετοιμασία αυτής της διάσκεψης του 2015 με τη συμμετοχή ε, της Προέδρου ε, και των Προέδρων των Τριών Επιτροπών και των ανώτερων ψηματούχων της Ρωσίας, της Αυστραλίας, της Ιαπωνίας, της Νότιας, της Νότιας Αφρικής και άλλων. Ευχαριστώ και αναμένω ε, τη συζήτηση. Mm, Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρέσβη. Περισσότερο δήλωση παρά ερώτηση. Πιστεύω ότι η πολιτική αυτή για τη μη διάδοση και την αναθεώρηση αυτής της συνθήκης αποτελεί μια συνενετική προσέγγιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι διαφέρουμε εδώ στο Κοινοβούλιο ή σε ό,τι αφορά τις κυβερνήσεις μας από αυτή την άποψη. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δώσουμε όλη μας τη στήριξη στους εκπροσώπους αυτούς που συμμετέχουν σε αυτή τη διάσκεψη, ξεκινώντας από τον είπα εκπρόσωπο. Ευχαριστώ κύριο Σκόν. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον ομιλητή μας. Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις. Θα ήθελα καταρχάς να αναφερθώ στο σέμα της Ινδίας και του Πακιστάν που θεωρείται ότι παίζουν καθοριστικό ρόλο στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Ξέρουμε ότι εκεί έλαβαν χώρα τρεις πόλεμοι. Ξέρουμε ότι το Κασμίρ έχει τη μεγαλύτερη, ε, το μεγαλύτερο αριθμό στρατευμάτων στον κόσμο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερο έτσι ώστε να διασφαλίσουμε το ότι δεν θα προκύψει ένας άλλος πόλεμος που θα οδηγήσει σε έναν άλλο σε ένα πυρηνικό πόλεμο μεταξύ αυτών των χωρών. Το δεύτερο, εδώ και λίγο καιρό βρισκόμαστε μάρτυρες των όσων συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή. Μία περιοχή πάρα πολύ ευαίσθητη που αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, προβλήματα με το Ιράν σχετικά με θέματα πυρηνικής, χρήση ε, όπλων. Πού ακριβώς έγκυται η δυσκολία στο να απαλλάξουμε από τα πυρηνικά όπλα ή από τα όπλα μαζικής περιοχής ε, καταστροφής όλη την περιοχή της Μέσης Ανατολής. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε έτσι ώστε να απαλλαγεί από όλα αυτά η Μέση Ανατολή. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δανόρντεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Σαφώς είμαστε υπέρ της μη διάδοσης των πυρηνικών και της διάσκεψης για την αναθεώρηση της συνθήκης. Θα πρέπει βεβαίω να έχουμε συνείδηση του πού έγκυται τα πραγματικά προβλήματα. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, έχουμε επανήλθε το θέμα της, του μονομερούς αφοπλισμού Υπάρχει μια ολόξυλη εκστρατεία στο Ηνωμένο Βασίλειο ε, σχετικά οικία θέματα από τη δεκαετία του 50 και του 60. Η Ρωσία, για παράδειγμα, που χρησιμοποιεί παρεμφερή πολιτικά όπλα σήμερα, απειλώντας χώρες με πυρηνικές επιθέσεις σε περίπτωση που δεν συμφωνήσουν με την ε, ρωσική πολιτική. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλές αναμνήσεις από το παρελθόν. Το δικό μου πρόβλημα είναι άλλοι φορείς και η δυνατότητα που έχουν να έχουν πρόσβαση σε μη σχάσιμο υλικό και στην τεχνοσγωσία που θα τους επιτρέψει να αναπτύξουν κάποιον εξοπλισμό, είτε πρόκειται για πυρηνικό όπλο ή για οποιοδήποτε άλλο όπλο. Μιλάμε για φορείς που δεν έχουν σχέση με κυβερνήσεις. Και αυτό βεβαίως θα είχε πολύ μεγάλες καταστροφικές επιπτώσεις αν βρεθεί σε λάθος χέρια Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά το αυτοβαστίγωμα είμαστε πάρα πολύ καλοί. Περνάμε το χρόνο μας στις δυτικές δημοκρατίες θέτοντας ερωτήματα στον εαυτό μας ενώ πραγματικά υπάρχουν αλλού πραγματικοί κίνδυνοι και απειλές που θα, όπου θα πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας και θα με ενδιέφερε να γνωρίζω την άποψή σας σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την επίλυση αυτών των θεμάτων. Το θέμα αυτό ετέθη από τον κύριο Κάνερ, το θέμα του Κασμίρα δηλαδή. Αν το Πακιστάν σταματήσει την αποστολή τρομοκρατών πέρα από τη γραμμή ελέγχου στην Ινδία και <clears throat> συνεχώς υποστηρίζει μια τόσο δύσκολη κατάσταση, τα πράγματα θα είναι πολύ λιγότερο απειλητικά. Και βεβαίως ένας από τους μεγαλύτερους υπέτειους ήταν ο Έουκιου Κάνο, ο οποίος ήταν υπεύθυνο για τα όσα συνέβησαν. Βεβαίως παράλληλα και το γεγονός ότι και το Ιράν βρίσκεται σε φάση ανάπτυξης πυρηνικών όπλων. Πιστεύω ότι το Πακιστάν είναι κατά ένα μεγάλο μέρος υπεύθυνο για όλα αυτά. Δεν θα ήθελα να ξεκινήσουμε μια συζήτηση για το Πακιστάν. Εσείς όμως θέσατε το θέμα του Κασμίρ. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σαμπάιος. Ευχαριστώ. Πιστεύω ότι η διεξαγωγή αυτή τη συζήτηση είναι πολύ σημαντική γιατί με αυτόν τον τρόπο έχουμε μια καθαρή εικόνα των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιμένω να βάλετε τα ακουστικά σας. Όπως έλεγα, είναι πολύ σημαντικό να επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτό το σημείο. Έχουμε 16.000 πυρηνικά όπλα σε όλο τον κόσμο και αυτός είναι ένας μείζον κίνδυνος. Υπάρχει και ο κίνδυνος βεβαίως ατυχήματος. Έχουμε ακούσει πολλά για το ατύχημα στη Φουκουσίμα. Γνωρίζουμε τις επιπτώσεις για την Ιαπωνία και τις παρακείμενες περιοχές. Και αυτές οι επιπτώσεις θα παραμείνουν για πολλές δεκαετίες ακόμα. Αυτός είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να προσμετρήσουμε τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις που έχει μια πυρηνική έκρηξη, ένα πυρηνικό ατύχημα. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή που επηρεάστηκε από το ατύχημα του Τσερνομπίλ. Ακόμα νιώθουμε τις επιπτώσεις αυτού του ατυχήματος. Ζω στη Σουηδία. Τι θα συμβεί ε, μετά από μια πυρηνική έκρηξη. Μια έκρηξη δεν επηρεάζει μόνο τις παρακείμενες περιοχές, μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές ανάλογα με τις βροχοπτώσεις. Θα πρέπει λοιπόν ε, να ασχοληθούμε περισσότερο με τις ανθρωπιστικές επιπτώσεις και θα πρέπει να βασίσουμε την επιχειρηματολογία μας σε τέτοιου είδους αίματα όταν μιλάμε για πυρηνικά όπλα. <clears throat> Ανθρωπιστικοί λοιπόν λόγοι. Ο κόσμος μας είναι λιγότερο ασφαλής από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Στο παρελθόν είχαμε τη βεβαιότητα ότι δεν θα χρησιμοποιούνται τα πυρηνικά όπλα. Υπάρχει τώρα ο κίνδυνος και υπάρχει ε, υποψία ότι κάποιος κάποτε θα, θα προσφύγει σε ένα πυρηνικό, ε, θα καταφύγει σε ένα πυρηνικό όπλο. Υπάρχει συμφωνία του Κοινοβουλίου σχετικά με, μια κοινή, με ένα κοινό ψήφισμα που στην ουσία... Αυτό είναι το δικό μας όραμα. Έτσι θέλουμε να συνεχιστούν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη διάσκεψη μη διάδοση πυρηνικών. Εγώ δεν έχω παρετηθεί ακόμα από την ιδέα ότι ενδεχομένω θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μία συμφωνία ή σε ένα ψήφισμα κυρίως γιατί δεν γνωρίζουμε κατά πόσον το Συμβούλιο θα καταλήξει σε μια κοινή θέση. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές απόψεις από πολλές διαφορετικές χώρες μετά την κρίση της Ουκρανίας. Τώρα η εικόνα έχει αλλάξει ριζικά. Δεν μιλάμε, ε, για εξοπλισμούς και όχι για αφοπλισμό. Από αυτή την άποψη η γνώμη του Κοινοβουλίου είναι ακόμα περισσότερο σημαντική. Αν μας φοβίζει η χρήση των πυρηνικών όπλων, τότε θα πρέπει να είμαστε απόλυτα ξεκάθαροι στην ε, άποψη που υιοθετούμε και θα πρέπει να στραφούμε και προς το Συμβούλιο και προς τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη σχετικά με αυτό το θέμα. Ξέρω ότι ο Κλάους, ε, ε, ο Επίπρος θα παραστεί σε αυτήν την συνάντηση μου ζήτησε να σας πω ότι τον απασχολεί ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν έχουμε καταλήξει σε μία συμφωνία. Έχουν υποβληθεί πολύ καλά ψηφίσματα. Υπήρξε ένα ε, ψήφισμα το 2010 με ένα άλλο το 2013. Δεν υπάρχει στην ουσία κάποιο πρόσκομα στην έκφραση των απόψεών μας κατά τη διάρκεια της διάσκεψης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καν θέλει να σχολιάσει την παρέμβαση του κύριου Φανόρντεν. Παρακαλώ. Να πω κάτι στον ε, συνάδελφο Τζέφρι. Είπα η Ινδία και το Πακιστάν και η δυσχέρεια σε σχέση με το Κασμία. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Μπορούμε να περάσουμε δύο ώρες να το συζητήσουμε. Είναι περίπλοκο το θέμα αυτό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό να μην απαντήσω σε αυτά που είπατε. Μπορούμε να συζητήσουμε για το πόσο έχει συμμετάσχει το Πακιστάν σε αυτές τις δραστηριότητες, αλλά επίσης μπορεί να ισχυριστεί κάποιος ότι και η Ινδία δεν είναι αθώα. Έχει παρέμβει στο Αφγανιστάν, στο Νεπάλ, στο Πακιστάν υποστηρίζει διάφορα αποσχιστικά κινήματα, πολλά παραδείγματα. Αλλά εγώ δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι χειρότερος από τους δυο. Εγώ ως ε, ενδιαφέρομαι να υπάρξει μια λύση για το θέμα αυτό με βάση το χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, τη χάρτα των Ηνωμένων Εθνών, ούτως ώστε οι κάτοικοι του Κασμίρ να αποφασίσουν τι θέλουν. Θα ήθελα να γίνει αυτό, γιατί είναι τρομερό τόσοι πόροι και τόσοι κίνδυνοι που υπάρχουν στο Πακιστάν, στο, στο Κασμίρ. Στην Ινδία υπάρχουν 55 εκατομμύρια, για παράδειγμα, φτωχοί που θα μπορούσαν να υποφεληθούν από αυτού του πόρου για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωή του και όχι για να σκοτώνονται. Και συνολικά θα ήθελα να αναπτυχθεί η Νότια Ασία. Όπως είδαμε στην Ένωση, μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερη πρόοδο, όχι μέσω πολέμων, αλλά μέσω συνεργασίας. Αυτή είναι η πρόθεσή μου και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε γι' αυτό. Ευχαριστώ κύριε Κάνη. Κυρία Βέλτμανς, λέει η πρόεδρος. Ευχαριστώ. Ήρθα λίγο αργά, αλλά ήμουνα σε κάποια άλλη επιτροπή. Ίσως ε, να ε, κάνω ερωτήσει, στις οποίες έχετε ήδη απαντήσει. Πριν από μερικά χρόνια πήγα στην Ιαπωνία. Πήγα στη Χειροσύμα και τον Αγκασάκη. Είδα τις, τα οδυνηρά κατάλοιπα σε αυτή τη χώρα. Άρα το βασικό, κατά τη γνώμη μου, είναι να συνεχίσουμε τον αγώνα για την απαγόρευση όλων των πυρηνικών όπλων και συμφωνώ πολύ με αυτά που είπατε αγαπητοί συνάδελφε να υπάρξει ένα ψήφισμα αλλά βέβαια ξέρω ότι πολλές φορές ε, τα ψηφίσματα του Κοινοβουλίου δεν έχουν συνέχεια αλλά θα ήταν ισχυρό μήνυμα αν μπορούσαμε να έχουμε ένα νέο ψήφισμα κατά τη διάρκεια της διάσκεψης για παράδειγμα στη Νέα Υόρκη τι θα γίνει όμως εκεί έχω το εξής ερώτημα Ποιο περιμένετε να είναι το αποτέλεσμα. Τι θα ήταν ικανοποιητικό αποτέλεσμα για σας. Βέβαια δεν θα αλλάξει ο κόσμος από τη μια στιγμή στην άλλη. Αλλά να υπάρξει κάποια πρόοδος. Και τώρα όταν κοιτάζω τον κόσμο, όταν βλέπω όλες τις σειράξεις, γίνομαι κάπως απεσιόδοξη. Βεβαίως ε, γίνονται βήματα αλλά προς τα πίσω. Τι περιμένετε λοιπόν, τι θα ήταν ικανοποιητικό ως αποτέλεσμα. Επίσης, οι περισσότερες χώρες που θα συμμετάσχουν σε αυτή τη διάσκεψη είναι δυτικές χώρες με τις δυτικές αξίες. Πώς θα πείσουμε τις χώρες λοιπόν της Μέσης Ανατολής να συμμετάσχουν, να βοηθήσουν να σημειωθεί η πρόοδος, να καταλήξουμε σε κοινό τρόπο σκέψης. Αυτό είναι μία από τις βασικές προκλήσεις. Τέλος. Γιατί λοιπόν να εγκαταλείψουν οι χώρες της Μέσης Ανατολής ένα ισχυρό μέσο που έχουν για να προωθήσουν τους στόχους τους. Πώς θα τις πείσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σαφχάουζαν. Ευχαριστώ. Πολύ σημαντική εργασία μπορεί να γίνει για τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων. Εισαγωγικά να τονίσω ότι όταν υπάρχει χρήση πυρηνικών όπλων υπάρχουν λόγοι. Όταν ε, οδηγήθηκαν οι Ηνωμένε Πολιτείε να ρίξουν ατομικές βόμβες, το έκαναν, γιατί θεωρούσαν ότι ήταν δίκαιος ο λόγος ήταν δίκαιο ο πόλεμος, άρα και δίκαια η χρήση των ατομικών όπλων. Βεβαίω η επιδίωξη της ειρήνη είναι πάντα δίκαιος στόχος. Εμείς βέβαια έχουμε κάπως μονομερείς απόψεις, δογματικές απόψεις, μη ισορροπημένε, προπαγανδιστικές. Αν έχουμε ξεχάσει την ε, διαδικασία για να βρούμε την αλήθεια. Αν, ξεχά, αν ξεχνάμε την ιστορία, στην ουσία ευνοούμε μακροπρόθεσμα τη χρήση των πυρηνικών όπλων. Γιατί μόνο αν πιστεύεις ότι εγώ έχω δίκιο, εγώ ξέρω την αλήθεια και άλλοι έχουν άδικο, μπορείς να πιστείς ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις πυρηνικά όπλα. Και έτσι μπαίνουμε σε μία οδό που θα μας οδηγήσει στη χρήση πυρηνικών όπλων. Θα πρέπει λοιπόν ευθύ εξ αρχής να ανησυχούμε πολύ περισσότερο για το ποιος έχει δίκιο, ποιος λέει την αλήθεια. Να μην παίρνουμε θέση υπέρ του α κατά του β, γιατί αυτό οπωσδήποτε θα μας οδηγήσει στον πόλεμο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Δεν υπάρχουν άλλοι ομιλητές. Οπότε να σχολιάσω κι εγώ. Κύριε Πρέσβη, παρά τα καθησυχαστικά λόγια του κυρίου Γκάλερ και τις αμφιβολίες της κυρίας Θεβάγιος, να σας κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Ποιες είναι οι θέσεις των κρατών μελών και τι ε, δυνατότητες διαβλέπετε να υπάρξει συμφωνία να καταλήξετε σε μια συντονισμένη θέση. Δεύτερον, πώς εκτιμάτε τις πρόσφατες ρωσικές δηλώσεις για το ενδεχόμενο της εισαγωγής πυρηνικών όπλων στην Κρυμαία. Δεν βοηθάει τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης κάτι τέτοιο. Είναι παραβίαση του υπομνήματος της Βουδαπέστης και οι μεταγενέστερες δηλώσεις της ε, Ρωσίας υπονομεύουν τις προσπάθειες ε, που έχουν γίνει για την προπαρασκευή της ε, συνδιάσκεψης αναθεώρησης, της REVCOM. Οι επιπτώσεις των διαπραγματεύσεων με το Ιράν για την ευρύτερη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. και τις πιθανότητες αφοπλισμού γιατί αυτή τη στιγμή είναι αντίθετη πορεία. Δημιουργείται τώρα ένα ΝΑΤΟ για την περιοχή του ε, κόλπου. Αυτά ως πρώτη δόση. Ευχαριστώ πολύ. Έχετε το λόγο κύριε Πρέσβη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ε, ευρωβουλευτές που έθεσαν μια σειρά από πολύ σημαντικά ζητήματα τα οποία θα επιχειρήσω να σχολιάσω με τη σειρά με την οποία ε, υπευλήθησαν. Ινδία, Πακιστάν πρώτα. Νομίζω ότι η πλειονότητα, αν όχι όλοι οι εμπειρογνώμονες επ' αυτού του θέματος θεωρούν ότι η ευρύτερη περιοχή Ινδίας-Πακιστάν είναι η περιοχή όπου ο κίνδυνος ε, πυρηνικής σύραξης από λάθος υπολογισμό είναι ο υψηλότερος στον κόσμο. Αυτό οφείλεται και στο ότι και οι δύο πυρηνικές δυνάμεις στην περιοχή αναπτύσσουν νέες δυνατότητες και από πλευράς όπλων, υποστρατηγικών και μέσω της δυνατότητας ε, χρήσης τους νέοι πύραυλοι δηλαδή αναπτύσσονται. Αυτό είναι οπωσδήποτε ιδιαίτερα ανησυχητικό. Και μας εκπλήσει ακόμη περισσότερο λόγω του ευρύτερου πλαισίου που αναφέρθηκε εδώ. Ότι είναι τόσο δεινή η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην ευρύτερη αυτή περιοχή. Αυτό το διαπιστώσαμε σαφέστατα και σε αυτά και στο μήνυμα του Πάπα Φραγκίσκου προς τη διάσκεψη της Βιέννης για τα πυρηνικά όπλα για το πόσο σπάταλες και άσκοπες είναι αυτές οι δαπάνες για πυρηνικά όπλα ενώ έχουμε τεράστιες οικονομικοκοινωνικές, οικονομικοκοινωνικές προκλήσεις. Κάτι άλλο που είπα την εισαγωγική μου ομιλία. Καλούμε όλα τα κράτη-μέλη να ενταχθούν στην ε, Συμφωνία για τη Μη Διάδοση ως μη πυρηνικά κράτη. Και φυσικά αντιτιθέμεθα και στις προσπάθειες υπονόμευσης της Συμφωνίας. Για να μην συμβεί αυτό, έχουμε ξεκινήσει ένα διάλογο και με την Ινδία και με το Πακιστάν για τη μη διάδοση, τον αφοπλισμό, αλλά και για θέματα πυρηνικής ασφάλειας και τους ε, προσφέρουμε βοήθεια. Θέτουμε στη διάθεσή τους βοήθεια. Ούτως ώστε οι ειρηνικές χρήσεις της πυρηνικής ενέργειας να γίνονται εφαρμόζοντας ε, τις βέλτιστες προδιαγραφές ασφαλείας, αλλά και διπλωματικά. Τους καλούμε να αξιοποιήσουν κάποια διεθνή μέσα. Για παράδειγμα, για μέτρα δημιουργίας κλίματος εμπιστοσύνης, όπως για παράδειγμα ο κώδικας ε, διοντολογίας της Χάγης για τη μη διάδοση βαλιστικών πυράβλων. Είναι ένα μέσο διαφάνειας για ανταλλαγή πληροφοριών, για ανταλλαγή ειδοποιήσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει πολύ αυτό τον κώδικα διοντολογίας. Τώρα, το επόμενο θέμα για τη RevCon, Θα υπάρξει ευρεία συμμετοχή θα συμμετάσχουν τα κράτη-μέλη σε μεγάλο βαθμό που ανήκουν, στην, που έχουν προσυπογράψει αυτήν την ε, σύμβαση. Οι αδέσμευτοι έχουν πολύ ισχυρή συμμετοχή. Και νομίζω ότι είναι καλό το επίπεδο διαλόγου μεταξύ όλων των ομάδων χωρών. Κάτι ιδιαίτερα σημαντικό που αναφέρθηκε από αρκετούς η ρωσική επιθετικότητα έναντι της Ουκρανίας και η παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας και η παραβίαση του υπομνήματος της Βουδαπέστης που είχε μια σειρά από διαβεβαιώσεις που είχαν δοθεί στην Ουκρανία το 1994 στα πλαίσια της ένταξης της Ουκρανίας στη διάσκεψη για τη, στην ε, σύμβαση για τη μη διάδοση ως μη πυρηνικό κράτος. Αυτό θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις για το μέλλον της μη και του αφοπλισμού συνολικά. Αν το συνδέσουμε μάλιστα και παραθέτω από αυτό που μόλις είπατε, μερικές από τις εμπριστικές δηλώσεις ε, της Ρωσίας που λέει ότι θα τεθούν σε κατάσταση συναγερμού κάποιες ρωσικές ε, πυρηνικές ε, δυνάμεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω είναι σαφής στη θέση της. Έχουμε καταδικάσει τη ρωσική επιθετικότητα, και το ότι έχουμε πει σαφώς ότι θεωρούμε ότι είναι παράνομη η προσάρτηση της Κρυμαίας και ελπίζουμε το θέμα της πυρηνικής ασφάλειας και των εγγυήσεων πυρηνικής ασφάλειας που πρέπει να δώσουν τα πυρηνικά όπλα προς τα, τα πυρηνικά κράτη, προς τα μη πυρηνικά κράτη και για να προωθήσουμε την ιδέα ε, ζωνών χωρίς πυρηνικά όπλα Ελπίζουμε λοιπόν όλα αυτά να μην υπονομευθούν από τις ρωσικές ενέργειες και να παραμείνουν στις προτεραιότητες όλων των κρατών όσον αφορά την πυρηνική ασφάλεια και την τρομοκρατία. Νομίζω ότι το ανέφερα στα 14 λεπτά της αγωγικής μου ομιλίας. Η πυρηνική ασφάλεια είναι ιδιαίτερα πρωταρχική προτεραιότητα για την Ένωση και είμαστε περήφανοι όχι μόνο γιατί συμμετέχουμε ενεργά στη διαδικασία που ε, ξεκίνησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε υπό την πρόεδρο Ομπάμα για την πυρηνική ασφάλεια, αλλά συμμετέχουμε και μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών μέσων. Ορισμένα είναι, για παράδειγμα, το Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά και μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας, όπου η Ένωση συμβάλλει στον προπολογισμό με 40 εκατομμύρια μεταξύ των κυρίων χρηματοδοτών του Ταμείου Πυρηνικής Ασφάλειας. Και χτυπάω ξύλο, αλλά μέχρι στιγμής η διεθνής κοινότητα έχει επιτύχει οι πυρηνικές δυνατότητες που υπάρχουν να μην πέσουν στα χέρια τρομοκρατών. Αλλά βέβαια το θέμα αυτό εξακολουθεί να είναι ύψιστη προτεραιότητα για όλους μας. Τώρα, τι θα επιτύχει αυτή η Ρευκόν. Είναι δύσκολο να είμαι πολύ συγκεκριμένος. Στα 14 λεπτά της εισαγωγικής μου ομιλίας, σε αυτά αναφερόμουν. Τι θα ήθελα να είναι η κατάληξη αυτής της ε, διάσκεψη. Θέλουμε να ενισχυθεί πρώτα απ' όλα η σύμβαση, να μην αποδυναμωθεί. Θέλουμε να υπάρξουν συμφωνίες για να σημειωθεί πρόοδος και για τους τρεις πυλώνες. Ίσως αυτή η πρόοδος ε, να μην είναι η καλύτερη, να μην είναι θεαματική, αλλά θα θέλαμε ουσιώδη. Τι σημαίνει να ενισχύσουμε την ε, συνθήκη αυτή ή τη σύμβαση. Δηλαδή να μην κάνουν και άλλες χώρες αυτό που έκανε η, Νότι... η, η Βόρεια Κορέα η οποία αποσύρθηκε από τη συνθήκη και άρχισε να κάνει πυρηνικές δοκιμές. Και θέλουμε να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι για το τι επιπτώσει θα έχει για μια χώρα εάν αποφασίσει να εφαρμόσει το άρθρο 10, δηλαδή το δικαίωμα απόσυρσης. Ότι θα υπήρχαν επιπτώσεις για την πυρηνική συνεργασία για αυτή τη χώρα και ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας των Εθνών θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το θέμα αυτό ως ενδεχόμενη απειλή προς τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια. Οπότε με αυτό περνάω στο θέμα της Μέσης Ανατολής και των κινήτρων. Τέθηκε ένα ερώτημα. Τι κίνητρα μπορούμε να προσφέρουμε. Τονίζουμε πρώτα απ' όλα την αρχή ότι αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να, να σπαστούν οι χώρες της περιοχής, να τη θεωρήσουν δική τους θα είχε έννοια μια διάσκεψη μόνο αν συμμετάσχουν όλα τα κράτη της περιοχής. Και η μερίσια διάταξη λοιπόν θα πρέπει να συμφωνηθεί μεταξύ των κρατών της περιοχής. Και άρα θα πρέπει να περιέχει κίνητρα για όλα τα κράτη για να έρθουν στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Πρέπει λοιπόν να δούμε το θέμα από μια σειρά πλευρές που υπάρχουν στην περιοχή. Μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Τι κίνητρα μπορούμε. Βέβαια, η κυρία είναι χαλεπή. Όλοι το αναγνωρίζουμε. Το περιβάλλον ασφάλειας αναφέραμε τι προβλήματα αντιμετωπίζει. Αλλά παρόλα αυτά, ακόμη και σε τέτοια περίοδο υπάρχει ε, περιθώριο πρόοδου. Για παράδειγμα, είχαμε τη διαδικασία αφαίρεσης των χημικών όπλων από τη Συρία. Μεγάλη επιτυχία παρά το ότι υπάρχουν ακόμη θέματα η Συρία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο στην ιστορία της περιοχής και σε καιρούς ιδιαίτερα έφλεκτους ενώ υπάρχει σύραξη, διεξάγεται σύραξη. Η Συριακή Δημοκρατία προσυπέγραψε την σύμβαση για τα χημικά όπλα και συμφώνησε να καταστραφούν τα χημικά της όπλα. Τη στήριξε πολύ γι' αυτό η Ένωση και τη στήριξε και συγκεκριμένα με 16 εκατομμύρια ευρώ. Άρα δεν θα πρέπει να χάνουμε την αισιοδοξία μας ακόμη και σε τόσο δύσκολες περιόδους όπως τώρα. Νομίζω ότι αν ε, ξαναδούμε τα κείμενα που ανέφερα στην αρχή της ομιλίας μου τη στρατηγική ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι εδώ εμείς στις Βρυξέλλες κατανοούμε τις προκλήσεις, τις απειλές και το πώς ε, συνδέονται αυτές οι απειλές. Αυτή η ανασφάλεια, η αστάθεια που υπάρχει στην περιοχή μπορεί φυσικά να δημιουργήσει ε, περισσότερη ζήτηση για αυτά τα όπλα μαζικής καταστροφής. Άρα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις τοπικές και περιφερειακές σειράξεις, τις κύριες. Το θέμα του Ιράν τέθηκε μια ερώτηση. Και η περιφερειακή του πλευρά από την Πρόεδρο. Αυτό είναι λίγο πέρα από τα θέματα της Ρευκών για τη διαπραγματεύσεις που προεδρεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση του 3 3 με το Ιράν στοχεύουν στην εξασφάλιση της αποκλειστικά ειρηνικής χρήσης της Ιρανικής πυρηνικής ενέργειας. και δεν ασχολούνται με το ενδεχόμενα στρατιωτικό παρελθόν αυτού του προγράμματος. Όπως είπα στην εισαγωγική μου ομιλία, έχει υπάρξει ήδη μια συμφωνία πλαίσιο και συνεχίζεται η εργασία και σε πολιτικό και σε επίπεδο πυρογνωμόνων για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία. Και αν γίνει αυτό θα έχει πολύ θετική επίπτωση στην ρευκόν και τις συζητήσεις της. Για το θέμα τώρα ενός ψηφίσματος του Κοινοβουλίου αυτό είναι δικό σας θέμα. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει ψηφίσματα για την συνθήκη μη διάδοσης και για άλλα θέματα που αντιμετωπίζει η υπηρεσία μας για τη συμφωνία για το εμπόριο όπλων και για άλλα σημαντικά θέματα που έχει εκφραστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να είμαι σαφής για να απαντήσω την ερώτηση για τη θέση της Ένωσης. Όλα όσα είπα στις παρατηρήσεις μου, χωρίς να προδικάζω την έκβαση, το πώς θα διαμορφωθούν δηλαδή τα πορίσματα του Συμβουλίου, όλα αυτά είναι στοιχεία της θέσης της Ένωσης για τη Ρευκόν. Η Ένωση και στη Γενική Συζήτηση αλλά και στις τρεις κύριες επιτροπές της Ρευκόν που θα ασχοληθούν με τη μη διάδοση, τον αφοπλισμό και τις ειρηνικές χρήσεις και ενδεχομένω και στα επικουρικά σώματα της Ρευκών εάν θα δημιουργηθούν ε, όταν θα αρχίσει η διάσκεψη που θα μπορούσαν να ασχοληθούν για παράδειγμα με περιφερειακά θέματα. Θέλουμε λοιπόν να συμμετάσχουμε σε όλα αυτά. Ευχαριστώ κύριε Σπρέσβη. Τα όσα είπατε μας οδηγούν στο τέλος της συζήτησής μας για την άποψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, επικείμενη διάσκεψη αναθεώρησης της συνθήκης στη Νέα Υόρκη. Ελπίζουμε να έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε εσάς και τους συνεργάτες σας μετά την, ε, το πέρας της συνεδρίασης και ελπίζω να πάνε όλα καλά κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων. Έχουμε αναποθέσει πολλές ελπίδες σε αυτή την άσκεψη, ενώ παράλληλα συνειδητοποιούμε ότι ζούμε σε εποχές πολλών προκλήσεων και ότι υπάρχουν πολλές απειλές για την κοινή μας ασφάλεια. Σας ευχαριστώ λοιπόν για τη σημερινή σας παρουσία. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ επιστρέψτε στις θέσεις σας. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησία διάταξη. Αφορά την έκθεση για τη στρατηγική, στρατιωτική κατάσταση στη λεκάνη της Μαύρης Θάλασσας μετά από την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας από τη Ρωσία. Ο εισηγητής είναι ο κύριος Ιωαν Μίρτσεα Πασκού και η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών αφού γίνει η πρώτη τους εξέταση είναι την 20, ήταν την 25η Μαρτίου γνωρίζω ότι ο κύριος Πασκού συναντήθηκε με πολλούς σκιώδεις εισηγητές και ελπίζω ότι επετεύθησαν αρκετοί συμβιβασμοί. Κύριε Πασκού, έχετε το λόγο. Well, Σας ευχαριστώ. Η έκθεση αυτή προσέλκυσε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δηλαδή που με θερμινεύτηκε σε 252 τροπολογίες. Χαίρομαι ιδιαίτερα. Οι μισές από αυτές τις τροπολογίες είναι πολύ καλές και θεωρώ ότι εμπλουτίζουν το κείμενο. Έλαβα υπόψη μου όλες τις τροπολογίες που θα μπορούσαν να συντελέσουν σε μια πληρέστερη έκθεση και κατέληξα σε 15 συμφωνίες, ε, τροπολογίες συμβιβασμού, τις οποίες συζήτησα χθε με μερικού από τους σκιώδες συζητητές. Το άλλο ίμιση των τροπολογιών είναι τροπολογίες που δεν μπορώ να δεχτώ, γιατί από τη μία πλευρά αμφισβητούν τα γεγονότα που αναφέρω στην έκθεση, θεωρώντας το μαύρο άσπρο, ή θέλουν να περιορίσουν το πεδίο, το εύρος της έκθεσης, κάτι που κατά την άποψή μου δεν είναι αποδεκτό. Χθε, όπως γνωρίζετε, συζητήσαμε το θέμα με τους συζητητές, τους υποβάλλουμε τις πρώτες 15 τροπολογίες συμβιβασμού. Έγινε μια συζήτηση, ε, ε, μπήκαν στο τραπέζι μερικές ιδέες για να ε, συμπληρωθεί αυτή η ομάδα των 15 τροπολογιών. Έγινε μια πρόταση για να γίνει αναφορά στην ε, τραντινιστερία υπερτινιστερία, γιατί ήταν ένα σχετικό θέμα. Μία άλλη πρόταση ήταν να, να εστιάσουμε την προσοχή μας περισσότερο σε θέματα πυρηνικών όπλων. Ένα ευαίσθητο θέμα ευαίσθητο όχι μόνο για αυτή την έκθεση αλλά γενικά στο Κοινοβούλιο είναι το είδος της υποστήριξης, της στήριξης που θα δοθεί σε στρατιωτικό επίπεδο στην Ουκρανία και εδώ αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε μια ορολογία που είχε υιοθετηθεί, τη διατύπωση που είχε υιοθετηθεί στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου για την Ουκρανία. Το άλλο, οι άλλες τροπολογίες θα προκύψουν αφού μετά από την προσεκτική ανάγνωση ε, του κειμένου από τους σχεδόν εισηγητές. Έχουμε προγραμματίσει μία άλλη συνάντηση την επόμενη εβδομάδα ή το αργότερο την εβδομάδα του Στρασβούργου και ζητήσαμε από τους κοιόδης συζητητές ε, μιλώντας τις ομάδες τους, αφού μιλήσουν τις ομάδες τους, να αποστείλουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο τις ε, προτάσεις, υποδείξεις που θα ήθελαν να κάνουν. Ένα πρόβλημα που είναι σημαντικό αφορά τη σχέση μεταξύ της συμφωνίας του ΜΙΣΚΑ και της έκθεσης. Ε, εάν γίνει μια αναφορά στη συμφωνία του Μίνς και για το συνδέσουμε την έκθεση μια κατάσταση που κινείται γοργά δεν νομίζω ότι θα καταφέρουμε και πάρα πολλά. Η αναφορά στη συμφωνία του Μίνσκ θα πρέπει να είναι γενική. Και θα πρέπει να σας πω ότι χθες μόνο Ε, ε, ρίχθηκαν 700 βλήματα κοντά στο αεροδρόμιο. Απλά και μόνο για να έχετε μία ιδέα. Ένα άλλο στοιχείο, υπάρχει ένα χωριό κοντά στη Μαριούπολη που λέγεται Σιρόκε, που είναι ένα μέρος όπου διεξάγονται πάρα πολύ σκληρές συγκρούσεις παρόλη τη συμφωνία του Μίσκα. Και βεβαίως οι ΜΕΝ ρίχνουν το βάρος τους ΔΕ για να μπορέσουν να δικαιολογήσουν τα όσα συμβαίνουν εκεί. Και ενδεχομένως στο μέλλον θα διαπιστώσουμε ότι η συμφωνία του ε, Μίνσκ δεν ισχύει, δεν εφαρμόζεται. Ελπίζω να μην συμβεί. Σε κάθε περίπτωση ε, θέλω να πω ότι το Μίνσκ δεν αναφέρεται άμεσα στην ουσία της έκθεσης. Θα ήθελα να σας παραθέσω δύο στοιχεία ακόμα. Ένα κομμάτι του Παλαισιανού αεροσκάφους απομακρύνθηκε από τους κατοίκους της περιοχής και δόθηκε στην ε, στην Ρωσία όσο τρόπεο, όσο τρόπεο και εκτίθεται ως τρόπεο. εκφράζοντας ε, την ευγνωμοσύνη για την στήριξη από ε, τον τόπιο πληθυσμό. Ένα άλλο θέμα που είναι ενδιαφέρον είναι ότι μετά από την συζήτηση ή μάλλον την απόφαση της Ρωσίας να πουλήσει S-13-300 στο Ιράν, ε, το Ισραήλ ανέφερε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο πώλησης ή παραχώρηση όπλων στους Ουκρανούς. Αυτό είναι ένα άλλο στοιχείο που έχει κάποια βαρύτητα. Όλα τα στοιχεία που παρατίθεται σε αυτή την έκθεση είναι τεκμηριωμένα πολλά προέρχονται από το ανώτατο αρχηγείο της Ρωσίας. Ε, ε, αναφέρεται ότι μετά από την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας η Ρωσία δημιούργησε μία δύναμη κρίση ε, στην Κρυμία, ε, Κρυμαία. Αυτοί που δεν θέλουν να δουν αυτή την πραγματικότητα θα πρέπει να πάνε στον ανώτατο αρχηγείο και να το επανεξετάσουν το θέμα. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους μου και ιδιαίτερα τους σκιώδεις εισηγητές για τη συνεργασία τους. Προσπαθούμε να ενσωματώσουμε όσο γίνεται περισσότερα στοιχεία, ακόμα και από συναδέλφους που ε, δεν, δεν θα δεν είχαμε σκεφτεί στην αρχή. Προσπαθούμε λοιπόν όλα αυτά να συμπεριλάβουμε στη Συμφωνία συμβουλισμού. Ευχαριστώ κύριε Πάσκο για τις προσπάθειές σας. Θα ήθελα τώρα να οργανωθούμε λιγάκι σε ό,τι αφορά τη συζήτηση. Κύριε Γκάλαρντ θα μιλήσει σε τεκμέρους του κύριου Λάνκμπεργκ, του σκιώδη συγητή του ΕΛΚ. Ναι, Μου ζήτησε ο κύριος Λαγκμπέργκερ να τον ε, αντικαταστήσω. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ευρεία συνένεση και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας. Έρχεται την κατάλληλη στιγμή και βεβαίως θα πρέπει και εμείς να τη συζητήσουμε. Πιστεύω ότι τα μηνύματα που στάλθηκαν από το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο στους ενδιαφερόμενους είναι μηνύματα σαφή, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ξεκάθαρη, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά αυτή την περιοχή. Ο συνάδελφος Λαντμπέργκερ είπε ε, ήθελε να αναφερθεί σε μια τροπολογία που δεν καλύπτεται από το συμβιβασμό. αναφέρθηκε σε μια παρεμφερή ε, εμπειρία των ε, ταγμάτων στην ε, Λιθουανία. Θα μπορούσε λοιπόν να εξεταστεί το ενδεχόμενο ενός κοινού τάγματος από θαλάσσις και ξυλάς και αυτό θα διευκόλυνε τον εξυγχρονισμό των αμυντικών δυνάμεων και θα αυξήσει και την δυνατότητα τις δυνατότητες στην Μαύρη Θάλασσα. Αυτό είναι ένα θέμα που δεν καλύφθηκε από τον, ε, τις συμβαστικές προτάσεις και μου ζήτησε να, τραβήξω, να ε, εστιάσω την προσοχή σας σε αυτό το σημείο. Θα ήθελα αυτά, ε, σας ευχαριστήσω για την συνεργασία. Galer, rozumiem, że pan Krasnodębski zastępuje sprawozdawcę cienia grup ECR, czyli Marka Jurka, tak? Bardzo proszę. Ε, κύριε ε, ο Μάριν Γιούρικ ε, είναι ο εισηγητής. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για τη θαυμάσια έκθεσή του. Οι συμβαστικές τροπολογίες, ότι καταλάβαμε δεν έχουν ακόμη διαμορφωθεί οριστικά, θα υποβληθούν λοιπόν. Ευχαριστώ γιατί πολλές από τις δικές μου τροπολογίες λήφθησαν υπόψη, ωστόσο να αναφερθώ σε ορισμένα άλλα θέματα επί των οποίων θα θέλαμε να παρακαλέσουμε να συμπεριληφθούν στις τροπολογίες. Το είπατε κι εσείς. Πρώτον, σε αυτή την έκθεση πρέπει να αναφερθούμε στα πυρηνικά όπλα. Το είπε και ο κύριος Γιούρεκ στην ομιλία του και συγκεκριμένα αναφέρθηκε στην τροπολογία 48. Ελπίζω να μπορέσουμε να βρούμε μια, μια, ένα συμβασμό επ' αυτού. Επίσης, θεωρώ ότι είναι σημαντικό να αναφέρουμε την υπερδνηστερία. Είναι μια περιοχή κλειδί για την ευρύτερη περιοχή. Και εδώ θέλω να βασιστώ στις τροπολογίες του κυρίου Γιούρεκ. Είναι οι τροπολογίες 135 και 138 και τελευταίο. Έχει γίνει μια έκκληση από τον πρόεδρο Ποροσέγκο για να υπάρξει μια ειρηνευτική αποστολή. Μήπως θα μπορούσαμε σε κάποιο σημείο να το αναφέρουμε και αυτό. Ξέρω ότι είναι δύσκολο να το βάλουμε στα πλαίσια της συμφωνίας Μίντς. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η εφαρμογή της. Και επίσης, κάτι που ίσως είναι λίγο ευρύτερο, αλλά εμείς ως Ευρωπαίοι θεωρούμε ότι από τη μία πλευρά υπάρχει ευρεία συμφωνία μεταξύ των διαφόρων πολιτικών ομάδων όσον αφορά τις σχέσεις, τις σχέσεις μας με τη Ρωσία αλλά ίσως τελικά να μην είναι τόσο ευρεία αυτή η συνένεση όσο ήταν στην περίπτωση της Γεωργίας όταν πριν από δύο χρόνια είχαμε αυτόν τον σύντομο πόλεμο αλλά παρά αυτήν την ε, ευρεία συνένεση. Πρέπει να πω ότι υπάρχουν σημαντικά ευρωπαϊκά κράτη που ακόμη υφίσταται τις επιπτώσεις λανθασμένων αποφάσεών τους στο παρελθόν. Για παράδειγμα, όπως ξέρετε έχουν ε, πουλήσει ε, ε, πολεμικά σκάφη τύπου Μιστράν στη Ρωσία. Ίσως πρέπει να το αναφέρουμε στην έκθεση αυτό. Και κάτι ακόμη. Πρόσφατα συζήτησα με έναν Πολωνό συνάδελφο, ο οποίος ε, ασχολείται πολύ με το θέμα της Ουκρανίας. Ήταν μία συνάδελφος και η, η, συνάδελφος αυτή με ενημέρωσε για κάτι που δεν είναι γνωστό στην κοινή γνώμη για τις φρικαλαιότητες που διαπράττονται από ό,τι φαίνεται γίνονται ε, μαζικοί ευνουχισμοί Ουκρανών νέων ε, κρατουμένων. Θα έπρεπε λοιπόν να εκφράσουμε την ανησυχία μας στην έκθεση αυτή και να τονίσουμε ότι πρέπει να τιμωρηθούν αυτά τα εγκλήματα. Για παράδειγμα, μέσω του Διεθνούς Δικαστηρίου της Χάγης. Σε κάποιο σημείο θα έπρεπε να το συμπεριλάβουμε σε αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Γενικά, Θα ήθελα να πω ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι πολύ σημαντική και είναι ένα πολύ καλός μηχανισμός αυτός που μας παρουσίασε ο συγητής και επαναλαμβάνω σε συντομία τα όσα είχα πει χθε στην συνεδρίαση των σκιωδών εισηγητών όσον αφορά ε, την ε, 6-11 ε, 3-6-11 και όσον αφορά την τροπολογία 153 που υπογραμμίζει την τουρκική πολιτική στη Μέση Ανατολή και όσον αφορά τον σημαντικό ρόλο της Τουρκίας στη Μέση Ανατολή, στην περιοχή αυτή και θα πρέπει πιστεύω να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στον εύξενο πόντο, στην περιοχή του ξενοπόντου και όχι ε, στην ε, νότια ακτή της Τουρκίας. Διότι θα μπορούσαν αυτά τα θέματα να ε, περιληφθούν στην έκθεση για την Τουρκία. Στον Συμβασμό 6 πάλι ή υπάρχουν αυτοί οι γεωγραφικοί περιορισμοί. Ε, ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αν αναφέρουμε τη Ρουμανία και την Πολωνία, παρόλο που η δεύτερη δεν είναι ακριβώς στον έξινο πόντο, θα πρέπει είτε να αποκλείσουμε την Πολωνία, είτε να περιληφθούν και οι χώρες της Βαλτικής που βρίσκονται στα όρια, ε, στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Ρωσία. Γενικά όμως δεν ξέρω πώς να λύσω αυτό το πρόβλημα. Ίσως ο εισηγητής μας προτείνει μια καλή λύση όπως κάνει συνήθως. Επίσης για το συμβασμό 11 και η τροπολογία του κ. Τένοκ ο οποίος προτείνει να δώσουμε στην Ουκρανία τα στρατιωτικά μέσα για να προσπίσει την επικράτειά της και η άλλη τροπολογία δεν είναι πολύ σαφής. Γι' αυτό παρακαλώ τον εισηγητή να χρησιμοποιήσει τη διατύπωση του ψηφίσματός μας για την Ουκρανία Τη 15 η Ιανουαρίου του 2015 και αν δεν απατώμε η γραμματεία ήδη κάνει αυτές τις κινήσεις. Για μία ακόμη φορά ε, είμαι πολύ ικανοποιημένο με αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Σατίνα. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας επί του γεγονότος ότι αυτή η έκθεση είναι εξαιρετική. Είναι μία έκθεση μεταξύ πολλών άλλων που συντάχθηκαν τους τελευταίους μήνες αρχίζοντας από την ε, Συμφωνία Σύνδεσης, την έκθεση Γκέις και αυτή η έκθεση δείχνει ότι ο εύξηνος πόντος είναι μία από τις πιο στρατηγικές ζώνες της εφηλίου. υπό την καθαρή έννοια της λέξης και υπό την ευρύτερη έννοια του όρου. Ε, στην ευρύτερη έννοια θα περιλαμβάνεται η Τσετσενία, τον Αργόνο Καραμπάκα, η Νότια Σωσετία και η Υπερδινιστερία. Αυτά είναι παραδείγματα προσπαθειών που καταβάλει η Ρωσία για να έχει το στρατηγικό έλεγχο του ευξήνου πόντου. Πριν από την κατοχή της Αυχαζίας, η Ρωσία δεν είχε λιμάνι στον εύξηνο πόντο, παρά στην ανατολική ακτή μία, δύο μικρά λιμάνια. Γι' αυτό το λόγο η Ρωσία προσπάθησε να ελέγχει ένα μεγαλύτερο λιμάνι, το οποίο και πέτυχε ε, με την Απχαζία. Λοιπόν, αυτή η έκθεση είναι καλή. Για ποιο λόγο. Επειδή ε, δείχνει ότι η Ευρώπη ενδιαφέρεται για την περιοχή του Ευξηνού Πόντου. Επειδή εάν σε σχέση με την Τσετσενία στην Αφχαζία στη δεκαετία του 90, όπου σε σχέση με την κατοχή της Αυγαζίας το 2008, εάν δεν θα είχαμε σιωπήσει, δεν θα είχε... Ε, ε, αν δεν είχαμε σιωπήσει δεν θα υπήρχε αυτή η προσάρτηση. Τώρα όμως λέμε σαφέστατα ότι πρέπει να δημιουργηθεί πάλι μια στρατηγική ισορροπία, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ισορροπία στην περιοχή. Αλλά η έκθεση υπογραμμίζει τα πιο σημαντικά, δηλαδή ότι πρέπει να καταδείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι να προασπίσουμε τις ευρωπαϊκές και ευρωατλαντικές αξίες μας. Γι' αυτό σας ευχαριστώ για τη σύνταξη αυτής της έκθεσης. Συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπατε. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνούμε λοιπόν όλοι. Ο κύριος Σαφχάουζερ. Ε, δεν μου αρέσει αυτή. Ε, ε, ε remarques. D'abord, δεν μου αρέσει αυτή η έκθεση, το φαντάζεστε. Δύο παρατηρήσει. Η πρώτη τεχνική φύσεω. Καταθέσαμε ορισμένε τροπολογίε. Δεν έχουμε ομάδε συνεπώ όχι σκιώδη εισηγητή. Αγαπητοί φίλοι, τίποτα δεν σα εμποδίζει να με καλέσετε. Νομίζω ότι από την αντιπαράθεση μπορεί να προκύψει μεγαλύτερη αλήθεια, τουλάχιστον από την αμοιβαία κατανόηση. Δεν μου αρέσει λοιπόν αυτή η έκθεση, επειδή είναι μία έκθεση μιας πλευράς, αν θέλετε, της δύση και όχι μια έκθεση ειρήνης. Δεν προσπαθεί να χτίσει γέφυρες δεν προσπαθεί κοντά ε, στη Δύση να δείξει τι αφορά σήμερα την Κίνα, την Ινδία, τη Βραζιλία, τη Ρωσία, έναν άλλο κόσμο. Ένα κόσμο όπου θα πρέπει να βρεθούν ισορροπίες. Δεν μου αρέσει λοιπόν αυτή η έκθεση επειδή κατά κάποιο τρόπο ζει σε ένα μη πραγματικό κόσμο. Δεν υπάρχουν από τη μία πλευρά δυνάμεις που αναζητούν τα συμφέροντά τους και άλλες που αναζητούν τα δικά τους συμφέροντα. Ζούμε σε έναν ε, κόσμο όπου μία μόνη δύναμη κάνει δηλώσεις και οι άλλοι πρέπει να ακολουθούν. Δεν μου αρέσει λοιπόν αυτή η έκθεση επειδή κατά κάποιο τρόπο είναι ανεύθυνη. Δεν λαμβάνει ε, υπόψη την πραγματικότητα. Θα ήθελα λοιπόν να επενθυμίσω, αγαπητέ φίλε, ορισμένα ε, γεγονότα. Ο κ. Κούγκαν αποφάσισε μετά από την 10η Σεπτεμβρίου να κάνει πόλεμο στο Ιράκ. Και τότε είπαμε ότι υπήρχαν όπλα μαζικής καταστροφής. Αυτό δεν ήταν η αλήθεια φυσικά. Υπήρχαν στρατηγικά συμφέροντα πίσω από αυτή τη δήλωση. Όταν η κυρία Νούλαν, η σύζυγος του κ. Κούμαν, δημιουργεί την ε, ε, Επανάσταση, δεν θα μου πείτε ότι είναι αυθόρμητες, ότι οφείλονται στη δημοκρατία, οργανώνονται κατευθύνονται, υποστηρίζονται οικονομικά. Αυτό σημαίνει ότι ζούμε σε μια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Και πιστεύω ότι η θέση της Ευρώπης δεν είναι να βρίσκεται στη μία πλευρά, αλλά να χτίζει γέφυρες, να προσπαθεί να βρίσκει ισορροπίες. Δεν πρέπει να εκπλαγείτε λοιπόν να ζείτε σε μια αντιπαράθεση. Και όσο πιο μικρή χώρα είναι και ποιος, μια χώρα είναι μικρή και θέλει τον πόλεμο, δεν πρέπει να επίσηστε όταν ζείτε σε μια λογική πολέμου που τελικά αυτή η λογική οδηγεί στον πόλεμο. Ο κ. Uh, uh, Ευχαριστώ. Καλή έκθεση γενικά. Αν ε, μπορώ να προσδιορίσω μία δυναμία είναι σε αυτά που λέει για την Τουρκία. Γιατί αν εξετάσουμε την περιοχή του Ευξήνου Πόντου, ποιο ελέγχει την είσοδο, στη μαύρη, την πρόσβαση στη Μαύρη Θάλασσα, ο ρόλος της Τουρκίας είναι ζωτική σημασία. Οπότε η Ευρωπαϊκή Ένωση ίσως θα έπρεπε να είναι πιο θετική, πιο ενθαρρυντική. Αντίθετα, στην έκθεση γίνεται παρόδο μια αναφορά στην Τουρκία, στην ιδεολογική σκέψη G και μερικοί από τους συνήθεις υπόπτους έχουν υποβάλει τροπολογίες που ε, συμπεριλαμβάνονται στην τρίτη συμβαστική που είναι πολύ πιο αρνητικές ε, προς την Τουρκία. Είναι τα συνήθεια αντιτουρκικά που ακούμε εδώ μέσα. Στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης είναι ιδιαίτερα λυπηρές τέτοιες αναφορές. Γιατί πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία είναι βασικός στρατηγικός εταίρος ιδιαίτερα για θέματα ευξήνου πόντου. Κατά τα άλλα είναι καλή έκθεση, στεναρή έκθεση και φυσικά αυτό ακριβώς περίμενα από έναν εισηγητή όπως ο πρώην ε, Ρουμάνος Υπουργός Άμυνας ε, συνάδελφος Πάσκου. Κάνει μερικές ευγενικές αναφορές στις ε, αντιδράσεις ε, ασφαλείας της Ένωσης. Υποθέτω ότι είστε υπογραμμένοι να το κάνετε, αλλά πολύ σωστά το κέντρο βάρους της εκθεσής σας τονίζει την ανάγκη να ενισχυθούν οι δυνατότητες δράσης του ΝΑΤΟ και ε, να αλλάξει η στάση του ΝΑΤΟ για την περιοχή. Έχει λοιπόν ε, εστίαση στο ΝΑΤΟ η έκθεσή σας. Να μην το ξεχνάμε αυτό. Για τα θέματα ασφαλείας το ΝΑΤΟ είναι ο κύριος ρόλος να μη μας ε, εκτρέψουν από το στόχο μας όλες αυτές οι ανοησίες για το ρόλο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Βέβαια καταλαβαίνω ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία και η Τουρκία είναι ε, σύμμαχοί μας στο ΝΑΤΟ και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος. Κύριε Γκάλερ θέλετε και πάλι να μιλήσετε. Ναι, να πω κάτι σύντομα για αυτά που είπε ο κ. Και εγώ είμαι υπέρ ενό πολυπολικού κόσμου. Δεν πρόκειται περί αυτού. Περί τίνο πρόκειται. Διευρύνει κανείς ε, την επιρροή του ει βάρο και κατά τη εκπεφρασμένη βούληση ενός ε, γειτονικού ε, έθνους. Αυτό είναι απαράδεκτο σε μια Ευρώπη του 21ου αιώνα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Ε, κύριε Γκάλερ, ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσω τον αγαπητό μου φίλο, τον κύριο Πάσκου, για τη θαυμάσια εκθεσή του. Γιατί η έκθεση με τις εξαιρετικές ε, και εκτεταμένες ε, συμβολές σας δείχνει κάτι που όλοι το περιμέναμε οι ενέργειες της Ρωσίας στην ε, Μαύρη Θάλασσα είναι τμήματα μια σταδιακής πολιτικής της Ρωσίας που τώρα περνάει σε κρίσιμη φάση με αυτήν την ε, επιθετικότητά της και την στάση προσπάθειας να επικρατήσει έναντι της Δύσης. Και υποθέτω ότι η Γαλλία εξακολουθεί να είναι δυτική χώρα ακόμη και για το Front National. Είμαι πεπισμένος ότι η Γαλλία έχει παίξει βασικό ρόλο για την ανάπτυξη της Δύσης. Δεύτερον, υπάρχουν πολλές ομοιότητες που αναφέρονται στην έκθεση μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Βαλτικής. τι εννοώ ομοιότητες. Και στις δύο παρατηρούμε ρωσική επιθετικότητα και στις δύο βλέπουμε ότι οι χώρες της περιοχής αισθάνονται εκτεθειμένες σε αυτήν την ε, επιθετικότητα. Τρίτον, βεβαίως η έκθεση σαφώς και εκπεφρασμένα λέει ότι η Ρωσία έχει μετατρέψει τη Μαύρη Θάλασσα σε προγεφύρωμα. Η Κρυμαία είναι οπλισμένοι μέχρι τα δόντια όπου έχουν εγκατασταθεί και τακτικά και στρατηγικά όπλα. Και το λέει επανειλημμένα η έκθεση. Αναφέρει τα τρία στοιχεία. Η, Ρώσα, η Ρωσία έχει αναπτύξει στρατεύματα, αεροσκάφη και πολεμικά ε, σκάφη που όχι απλώς αλλάζουν, έχουν εντελώς ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Το άλλο. Λόγω αυτών των ενεργειών της Ρωσίας, το ΝΑΤΟ για να συμμορφωθεί στις υποχρεώσεις και τα καθήκοντά του, είναι υποχρεωμένο να αντιδράσει, αναπτύσσοντας κάποιες περιορισμένες δυνατότητες ε, ανδρών και άλλων τακτικών όπλων, αλλά καμία σχέση με τον αριθμό που έχουν αναπτύξει στρατευμάτων και όπλων που έχουν αναπτύξει οι Ρώσοι. Και αυτό το λέει σαφώς η έκθεση. Αυτό, όπως ε, μας είπε ο θαυμάσιος γνώστης ε, κύριος Βαν Όρντεν, το ΝΑΤΟ είναι αυτό στο οποίο θα πρέπει να στραφούμε σε αυτή την περιοχή αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τη ρωσική επιθετικότητα. Η μόνη μας δυνατότητα ε, να αντιδράσουμε είναι το ΝΑΤΟ, είτε μας αρέσει είτε όχι. Κάτι άλλο που επίσης αναφέρεται στην έκθεση είναι ότι σε όλη την περιοχή αυτή διαπιστώνουμε εντυπωσιακή ρωσική προπαγάνδα που έχει το ρόλο της σε αυτόν τον υβριδικό πόλεμο που προωθεί η Ρωσία και μάλιστα με ιδιαίτερα επεξεργασμένο τρόπο. Άρα πρέπει να υπάρξει αντίδραση από πλευράς μας και η ύπατη εκπρόσωπος θα μας προτείνει προσεχώς μια κοινή προσέγγιση για να αντιπαρατεθούμε σε αυτή τη ρωσική προπαγάνδα. Ξέρετε ακόμη και τα πολιτικά κόμματα εδώ πληρώνονται από τη Ρωσία. Θυμάμαι τα πόσα SMS απεκάλυψε η εφημερίδα Le μεταξύ της Ρωσίας και των γραφείων ε, κάποιου πολιτικού κόμματος στο Παρίσι για να ευλογήσουν την ρωσική κατοχή. Και είναι επίσης τραγικά επίκαιρη αυτή η έκθεση. Διότι είναι ακτινογραφία εξελίξεων εμπορία που για να αντιμετωπιστούν χρειάζεται στρατηγική τροποποίηση των σχέσεων της Ένωσης με τη Ρωσία και τώρα και στο μέλλον. Γι' αυτό είναι ιδιαίτερα σκόπιμη η έκθεση του κυρίου Πάσχου και ο ρόλος της Επιτροπής μας είναι επίσης πολύ σημαντικός και θα συμβάλλουμε ουσιοδός στο να αλλάξει πορεία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέσω ακριβώς της ε, εποπτείας που ασκούμε στην ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική. Κύριε Σαφχάζερ, σέβομαι τους ε, κοινοβουλευτικούς κανόνες και πρόκειται να σας δώσω το λόγο, αλλά πριν το κάνω, σας παρακαλώ, τους πολίτες της περιοχής μου να τους αντιμετωπίζετε ισοτήμως, ως ισότιμους πολίτες και ισότιμους κοινωνούς του δυτικού πολιτισμού. Αυτό σημαίνει ότι και οι Ουκρανοί πολίτες. Εγώ εκπροσωπώ τους Πολωνούς. Είμαστε λίγο, λίγο πιο τυχεροί στην ε, ιστορία μας γιατί έχουμε την τύχη να είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν συμβούν όλα αυτά. Παρά το ότι εδώ και πολλά χρόνια είχαμε ήδη παρατηρήσει τις ε, λυπηρές εξελίξεις εντό της Ρωσικής Ομοσπονδίας και είχαμε προειδοποιήσει. Αλλά δεν μας άκουσαν. Αλλά δεν θα θέλαμε να μας αντιμετωπίζουν ως ε, χώρο αντιπαραθέσεων και ως χώρο επιρροής άλλων. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Δεν θα ήθελα να επισέλθω σε αυτό το θέμα. Θα ήθελα να θυμίσω ότι η τελευταία επίσκεψη η Κονολέσκη δημιούργησε πολλές, προβλήματα στις χώρες σας. Καταλαβαίνω το λόγο, λαμβάνοντας υπόψη τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισε η Ουκρανία τους Πολωνούς. Θα ήθελα να απαντήσω σε ό,τι αφορά τρία σημεία. Πολιτική της Γαλλίας. Η πολιτική της Γαλλίας βασίστηκε ε, ξεκίνησε από το στρατηγό Ντεγκόλ. Ο στρατηγός Ντεγκόλ ήταν ο πρώτος που διαπραγματεύτηκε με την Σοβιετική Ρωσία την εποχή εκείνη και με την κομμουνιστική Κίνα γιατί θεωρούσε ο Ντεγκόλ ότι η ισορροπία της ειρήνης απαιτεί ένα πολυπολικό κόσμο. Η πολιτική της Γαλλίας ελπίζω το μέλλον και πέρα από τους διάφορες διαιρέσεις θα παραμείνει αυτή μια πυρηνική δύναμη που επιθυμεί την ισορροπία της ειρήνης και όχι ενός στρατόπεδου. Γι' αυτό το λόγο ε, βγήκε η Γαλλία από το ΝΑΤΟ και ζητάμε την έξοδο της Γαλλίας από το ΝΑΤΟ και θα το εφαρμόσουμε αυτό. Το θέμα της ισορροπίας, ε, για να επανέλθω στη σημαντική έκφραση που χρησιμοποιήθηκε, ισορροπία, θα ήθελα να επανέλθω και πάλι σε αυτό το θέμα την πτώση του, μετά την πτώση του τείχους ακούστηκε και δεν είναι ψέματα. Υπάρχει ο καγκελάριος Κόλ ο οποίος διαβεβαιώνει ότι συμφωνήθηκε να μην υπάρξει διεύρυνση του ΝΑΤΟ και υπήρχε η πολιτική του αντί της αντιπυραυλικής ασπίδας στην Πολωνία που μας οδήγησε σε μία αντιπαράθεση μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προπαγάνδα, επιτρέψτε μου να πω ότι η Ρωσία είναι εκείνη ε, που δεν ε, εφαρμόζει το soft power. Εμείς είμαστε εκείνοι που ακολουθούμε την πολιτική του soft power και των ψεμάτων. Θα έλεγα ότι από τη δική μου άποψη τα πράγματα έχουν έτσι. Σε ό,τι αφορά την Κρυμαία, είχα την ευκαιρία να πω σε μία εφημερίδα ότι η Μαρή Λεπέν ήταν σαφώς αντίθετη στο να εμπλακούμε εμπισήμως στην διαδικασία αναγνώρισης της Κρυμαίας. Παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε την αναγνώριση της Κρυμαίας όταν έγιναν εκλογές στη χώρα. Θα ήθελα να πω παρόλα αυτά ότι δεν θέλουμε να εφαρμόσουμε την πολιτική των δύο μέτρων και δύο σταθμών. Το... Αυτό που δεχτήκαμε στο Κωσυφοπέδιο το αρνούμεθα στην Κρυμαία. Υπάρχει μια αρχή διεθνούς δικαίου για το δικαίωμα αυτοδιάθεσης των λαών ανεξάρτητα από το καθεστώς. Αν αύριο γίνουν ε, εκλογές, η Κρυμαία θα επιλέξει την προσάρτηση, ή την επιστροφή στη Ρωσία. Αυτό είναι ένα δημοκρατικό γεγονός που δεν αφισβητεί κανείς ούτε καν οι Αμερικάνοι. Η άποψή σας, η άποψη του Κοινοβουλίου είναι πολύ λιγότερο εξισορροπισμένη από αυτή της ε, ε, ε Γνωρίζουμε ότι ποτέ δεν θα επανέλθει στην Ουκρανία. Καταλαβαίνω ότι δεν ήσασταν παρόν καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης όταν οι καλεσμένοι μας παρέθεσαν τις απόψεις τους σχετικά με την κατάσταση της Κρυμαίας και του λαού της Κρυμαίας και το πώς συνέβαλαν στην ιστορία της Κρυμαίας καθώς και σε ό,τι αφορά τη δική τους άποψη σχετικά με την επιστροφή της Κρυμαίας στη Ρωσία. Ήταν ριζικά αντίθετοι και έχουν μία ξεκάθαρη άποψη. Ο κύριος Πασκού, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω μια προσπάθεια να απαντήσω εντάχει σε όλα τα σημεία που αναφέρθηκαν. Πυρηνικά όπλα Ναι, θα γίνει η μνήα αυτού του θέματος, το συμφωνήσαμε χθε. Αναφέρθηκα σε αυτούς σε αυτές τις συγκρούσεις που γίνονται σε αυτή την περιοχή, σε αυτή τη λεκάνη. Δηλαδή αναφέρθηκα σε όλα τα θέματα που θίξατε η αναγνώριση, μη αναγνώριση των συνθήκων που υπέγραψε η Ρωσία με την ε, Αυγασία και την Νότιο Σωτία επίσης αναφέρονται εδώ. Θα δούμε τι θα μπορούσαμε να βάλουμε, να συμπεριλάβουμε εδώ. Κύριε ναι, θα γίνει μία αναφορά στην Βαλτική. Γιατί μιλάμε για όλη τη γραμμή, δεν περιοριζόμαστε γεωγραφικά. Η υποστήριξη προς την Ουκρανία θα συμπεριληφθεί στο ψήφισμα που ανέφερα. Όταν αναφέρθηκα στη στρατηγική ισορροπία, ενδεχομένως τα αγγλικά δεν είναι και τόσο σωστά, είπα ισορροπία υπερισ της περιοχής της Μαύρης Τάρασσας. Δεν είναι μέσα στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν θέματα εκτός της περιοχής που θα χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση που προκύψει κάτι στην ε, περιοχή. Συμφωνώ ότι οι απαντήσεις που δώσαμε σε μερικές επιμέρους ε, κρίσεις ενδεχομένως μας οδήγησαν στην αντιμετώπιση ενός μείζωνος προβλήματος σαν την Ουκρανία. Αυτό είναι κάτι που αναφέρθηκε στην έκθεση τώρα. Θα δούμε τώρα το θέμα της ε, Τουρκίας και της επικοδομητικής προσέγγισης. Ξέρετε ότι έλαβα μία επιστολή από τον Τούρκο πρεσβευτή στην οποία επιστολή θέτει τέσσερα σημεία. Δύο σημεία είναι αποδεκτά. Τα άλλα δύο δεν είναι αποδεκτά. Ε, ένα από αυτά είναι ότι θα πρέπει να αντικαταστήσει τη λέξη Βόσπορους με τα ασθενά της Τουρκίας. Ε, του είπα ότι έχω να κάνουμε με γεωγραφικούς όρους και όχι πολιτικούς όρους. Θα σας δώσω το λόγο, περιμένετε. Ναι, ναι, είπα ότι προσπαθούμε να είμαστε επικοδομητικοί, αλλά όχι και υπερβολικά επικοδομητικοί από αυτή την άποψη. Κύριε Βανόρντερ, πιστεύω ότι για την αντιμετώπιση αυτού του υβριδικού πολέμου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει περισσότερα μέσα στη διάθεσή της πολιτικά μέσα και εδώ ξέρετε ότι θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι και θα... σε κάθε περίπτωση αυτή είναι μια μακρά συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Γκάλατ, κύριε Ποστινάρου, κύριε Γκάλατ. Ναι, τέτοιο αυτό το θέμα από τον κύριο Λανσμπέργη. Θα ήταν ευκταίο να υπάρχει μια στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των τριών αυτών χωρών. Αλλά αν μιλάμε μόνο για ένα τάγμα, αυτό είναι ασήμαντο. Ναι, κάτι τέτοιο, ένα τάγμα δεν αλλάζει και πολύ τα πράγματα. Κύριε Σαφχάουζε, σας επεφύλαξα τις τελευταίες μου παρατηρήσεις. Είπατε ότι η έκθεση αυτή είναι ανεύθυνη, επιτρέψτε μου να μην το σχολιάσω. Υπάρχουν πολλοί που δέχτηκαν αυτή την έκθεση, συμφώνησαν, δεν είναι ανεύθυνοι άνθρωποι θεωρήσατε ότι τουλάχιστον μερικοί από αυτούς είναι υπεύθυνοι. Είπατε ότι παρουσιάζω μόνο μία οπτική γωνία και εμέσως αφήνεται να εννοηθεί ότι δεν αναφέρομαι στη ρωσική πλευρά. Πραγματικά δυσκολεύομαι να βρω πού βρίσκεται η ουσία και πού βρίσκεται η προπαγάνδα και τι είναι αυτός ο ιδρυτικός πόλεμος. Γιατί σε τελική ανάλυση εδώ έχουμε μία παραβίαση διεθνούς δικαίου. Η μία πλευρά κάνει αυτό. Η άλλη πλευρά αντιδρά σε αυτό, την απόσπαση αυτού του κομματιού της χώρας. Εάν εγώ αναφερθώ και στην άλλη πλευρά, στη ρωσική πλευρά, θα το κάνω μόνο αναφερόμενο στα κίνητρα για την ε, παραβίαση του νόμου, που σε κάθε περίπτωση είναι κάτι απαράδεκτο. Γιατί αν το δεχτούμε εδώ, τότε δίνουμε το πράσινο φως σε όλους να το κάνουν. Ένα άλλο στοιχείο, Κωσίφτο, η Πορτογαλή Επανάσταση, ε, το Ιράκ. Ναι, ο στο Ιράκ. Το θέμα είναι, το κάνανε οι Αμερικανοί, γιατί να μην κλείσουμε τα μάτια μας αυτό που κάνουν οι Ρώσοι. Στην ουσία αυτή είναι η ουσία του επιχειρήματος. Που το ε, έγινε δεκτό από τους Αμερικανούς, ας το δεχτούμε και τους Όχι, όχι. Από την άλλη πλευρά είναι αμφισβητήσιμο ο ρόλος των Αμερικάνων και των χειρισμών στην Πορτοκαλία Επανάσταση κτλ. Ένα άλλο στοιχείο, ένα άλλο θέμα. Είπατε ότι αν ε, είμαστε επιθετικοί θα ε, οδηγηθούμε σε μια κλιμάκωση, ο πόλεμος θα φέρει πόλεμο κτλ λέτε ότι οι Ρώσοι πήραν αυτό που ήθελαν και τώρα θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Διαφορετικά θα ξεσπάσει πόλεμος αυτό, λέτε. Είναι αποδεκτό αυτό το επιχείρημα, πέστε μου, πέστε μου. Όχι, αυτό είπατε εμέσως. Γιατί είμαστε τόσο επιθετικοί στο, ε, σε ό,τι αφορά τα όσα έκανε η Ρωσία. Γιατί είμαστε τόσο επιθετικοί. θα το εξηγήσετε κάποια άλλη στιγμή. Νομίζω, ε, ή μάλλον αυτό μου θυμίζει ένα βιβλίο που εκδόθηκε στο τέλος της δεκαετίας του 50 ήταν του Πίτερ ε, Ουστίνοφ. Είχε φωτογραφίες και τίτλους. Έκανε ε, ότι ήταν ε, ο ε, πρέσβης διαφόρων χωρών. Σε μία περίπτωση είχε τον Κινέζο πρέσβη, ο οποίος έλεγε «Ο δράκος έξω από το σπίτι μας είναι καλύτερος από το κουνούπι μέσα στο σπίτι μας». Γιατί, και αυτός είναι ο λόγος απο το κουνουπι μεσα στο σπιτι μας επιτέθηκα στη Φορμόζα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε, αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα τη ρωσική προπαγάνδα ή τα ρωσικά κίνητρα, θα πρέπει να πούμε ότι η Ρωσία το έκανε αυτό και το λέω και το επαναλαμβάνω. Η, ωραία κοιμωμένη που ήταν το ΝΑΤΟ ξύπνησε μετά από το φιλί του πρίγκιπα, την Κρυμαία δηλαδή. Τώρα ο κύριος Πούτιν ε, ενοχλείται που η ωραία κοιμωμένη έχει θυμώσει. Εκείνος την ξύπνησε. Βρισκόμασταν σε μια δύσκολη θέση. Τι να κάνουμε με τον Άτο μετά το Αφγανιστάν. Είπε μισό λεπτό. Εδώ είμαι εγώ. Εδώ είμαι εγώ. Θα ασχοληθώ. Και ασχολήθηκε. Γιατί λοιπόν αυτό μας ενοχλεί. Το γεγονός ότι ξύπνησε η ωραία κοιμωμένη, αλλά ότι είναι θυμωμένη. Θα μπορούσε εύκολα να αποφευθεί αυτή η κατάσταση. Θα μπορούσατε να πείτε ότι ε, προσεγγίζει ο Ευρωπαϊκός στρατός δίχως την Κρυμαία, το ΝΑΤΟ θα ήταν εκεί που βρίσκεται. Περί αυτού πρόκειται το προκαλούμε και μετά κρίνουμε την αντίδραση στην ε, πρόκληση. Ξεχνιέται η πρόκληση, κρίνουμε την αντίδραση. Αυτό δεν είναι αποδεκτό, δεν είναι αποδεκτό με βάση τη λογική. Χαίρομαι ιδιαίτερα το γεγονός ότι δεν κάνατε άμεση επίθεση σε μένα ως άτομο. Απλά και μόνο δεν σας άρεσε η έκθεσή μου. Θα ήθελα να πω στους παρόντες και στους απόντες ότι μπορείτε να έχετε στη διάθεσή σας όλο τον κατάλογο των τροπολογιών, σαν να ήσασταν μέρος της όλης διαδικασίας, έτσι ώστε να ξέρετε ότι έτσι κινούμεθα. Υπάρχουν τροπολογίες, λάβαμε υπόψη τις τροπολογίες και θα πρέπει να σας ενημερώνουμε για τα όσα συμβαίνουν ε, σε ό,τι αφορά αυτή την έκθεση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Είχε ο επόμενο προσκεκλημένο μα, αλλά θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Βανχόρν. Κάτι θέλει να πει, όχι. Εντάξει. Ο κύριο Σαφχάουζε θέλει κάτι να πει, όχι. The vote on the report uh, takes... Η ψηφοφορία για την έκθεση θα γίνει στις 5 Μαΐου στην ΑΦΕΤ. Ευχαριστώ πολύ για μία ακόμη φορά κύριε Πασκού για τη θαυμάσια έκθεση. Ερχόμαστε τώρα στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Η ικανότητα ταχείας αντίδρασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε τον Γενικό Διευθυντή του Στρατηγικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον αντιστράτογο Βόλφκαμ Βόσολζομπε. Καλώς ορίσατε. Κύριε Στρατηγέ, παρακαλώ να μας ενημερώσετε σχετικά. Έχετε το λόγο. Thank you. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Διακεκριμένα μέλη του Προεδρού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ευχαριστώ που με προσκαλέσατε εδώ για να σας μιλήσω για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η στρατηγική αντίδραση και που βρίσκονται συζητήσεις όσον αφορά την στρατηγική πτυχή της ε, αμυντικής πολιτικής και πολιτικής άμυνας. Θα ήθελα, εάν συμφωνείτε, να σας παρουσιάσω ορισμένα βασικά στοιχεία του θέματος, δηλαδή τις ταχείας αντίδρασης γενικά, και κατόπιν θα ακούσω τις ερωτήσεις σας. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, ποια είναι η φύση ε, της στρατιωτικής αντίδρασης ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι μάχημες μονάδες αποτελούν το επίκεντρο, αλλά και πολλά περισσότερα αυτό το θέμα είναι πιο περίπλοκο. Βεβαίως χρειάζεται ένα κατάλληλο σύστημα διοίκησης και ελέγχου από το πολιτικό και στρατικό επίπεδο στο στρατικό επίπεδο φτάνοντας στις ε, μάχημες μονάδες. Κατόπιν χρειάζεται ένα, μια γρήγορη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Επίσης, έγκαιρη προειδοποίηση για να προετοιμαστεί η μάχημη μονάδα. Η Άγγελ προειδοποίηση βασίζεται στις πληροφορίες και στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βασίζεται ε, στις πληροφορίες που θα δώσουν τα κράτη-μέλη. Επίσης, χρειάζεται να προετοιμάσουμε το έδαφος για τη χρήση των μάχημων μονάδων με πολλές πολιτικές πληροφορίες και γνώσεις όσον αφορά ε, τους φορείς λήψεων των αποφάσεων σε πολιτικό επίπεδο. Τι είναι όμως μια μάχημη μονάδα από τεχνική άποψη. Καταρχήν, η μάχημη μονάδα, battle group, είναι μια ε, δύναμη κρούσης που περσέ δεν έχει καμία σχέση με την ταχύ αντίδραση, αλλά ε, έτσι περιγράφεται από τον ΝΑΤΟ. Δεν έχει απαραίτητο σχέση με τη μάχη. Έχει πολλαπλούς στόχους και στα πλαίσια Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα φτάσει στο υψηλότερο το επίπεδο της στρατιωτικής χρήσης. Ποιο είναι το μέγεθος αυτών των μονάδων. Αυτή τη στιγμή Έχουμε ένα ε, καλό παράδειγμα, το ε, βόρειο των σκανδιναβικών χωρών, της Σουηδίας δηλαδή, που περιλαμβάνει έξι χώρες και αποτελείται από ε, πεζικό, από μηχανοκίνητα οχήματα και έχουμε ε, αρκετές αρκετά μέσα όσον αφορά την επιτήρηση και την αναγνώριση. Και επίσης, εδώ έχουμε ε, μία γεωμορφία της Σουηδίας, έχουμε ε, μία αεροπορική πλευρά. Δηλαδή, υπάρχει μία κοινή μονάδα αυτή η αεροπορική πλευρά ε, περιλαμβάνει τακτικές μεταφορές, στρατηγικές μεταφορές και επίσης μαχητικά αεροσκάφη. Για να σας υπενθυμίσω το χρονικό διάγραμμα που καλύπτουν αυτές οι ε, μάχημες μονάδες. Όταν μιλάμε για τις... τη πιο στενό χρονικό περιθώριο, 15 μέρες από την προετοιμασία μέχρι την παρουσία των στατικών δυνάμεων ε, στο πεδίο των επιχειρήσεων, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι η διαδικασία προς τα άνω, δηλαδή ε, την έννοια τη διαχείριση της κρίσης, δεν έχουν περιορισμένο χρονικό περιθώριο, δεν είναι προκαθορισμένα. Έχουν διαδικασίες fast track, αλλά και αυτές οι γρήγορες διαδικασίες περιλαμβάνουν ποιες διαδικασίες χρειάζονται απολύτως, αλλά όχι τη διάρκεια αυτών μεταξύ της έννοιας της διαχείρισης κρίσης και της ε, απόφασης να ξεκινήσει επιχείρηση που λαμβάνεται από το Συμβούλιο θα πρέπει να γίνει επιχειρησιακό σχέδιο και θα πρέπει να είναι σε τιμότητα οι δυνάμεις μας. Και αυτό είναι δυνατόν με τις μάχημες μονάδες. Υπάρχουν και πιο στενά περιθώρια στο ΝΑΤΟ με τις Spearhead Forces, όπου προβλέπεται ότι θα υπάρχουν τρεις μέρες μόνο προειδοποίησης για να τεθεί σε λειτουργία η μάχη μονάδα. Το γεγονός ότι έχουμε πέντε ή τρεις μέρες προειδοποίηση, αυτό ε, ενέχει ένα παράγοντα κόστους για τα κράτη-μέλη. Κατόπιν έχουμε δέκα μέρες από την απόφαση να ξεκινήσουν την επιχείρηση μέχρι την έναρξη της επιχείρησης. Πάλι αυτό το χρονικό περιθώριο είναι πολύ πιεστικό. Τώρα θα ήθελα να τονίσω ότι η χρήση των μάχημων μονάδων θα έχουν επιτυχία αν υποστηρίζονται από μια γρήγορη πολιτική απόφαση. Εάν χρειαστεί πολύς χρόνος για να αποφασίσουν σε πολιτικό επίπεδο η υπεύθυνοι και μετά απαιτούμε γρήγορη ανάπτυξη των πολεμικών μέσων, πιθανόν δεν θα είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε ναι. σε επίγουσες καταστάσεις στο πεδίο των επιχειρήσεων. Και κατά κάποιο τρόπο έχουμε ένα καλό παράδειγμα εδώ για μια γρήγορη διαδικασία των αποφάσεων για την προετοιμασία ε, που έγινε στην ε, Κεντρική Αφρική. Τότε όμως δεν ακολουθήθηκε από τη χρήση μιας μάχημης μονάδας και η σύγκριση μεταξύ των ιδανικών χρονικών περιθωρίων και το χρόνο που χρειάστηκε ήταν 18 ε, μέρες. Δηλαδή ο χρόνος που χρειάστηκε από την απόφαση για να ξεκινήσει η διαχείριση χρήσεως μέχρι την άφηξη στο πεδίο των επιχειρήσεων ήταν 80 μέρες. Θα ήθελα να τονίσω ότι το παράδειγμα της ε, κεντροαφρικανής δημοκρατίας μας δείχνει ότι γρήγορες πολιτικές αποφάσεις είναι πιθανές και δυνατές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πέραν αυτού, επίσης, ε, ο, σχεδιασμός, ο μα σχεδιασμός μας περιλάμβανε τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, λιγότερο και από πέντε μέρες σε αυτή την περίπτωση. Επίσης, υπογραμμίζω τα πλεονεκτήματα που έχουν οι μάχημες μονάδες που δεν έχουν σχέση με την ταχύ αντίδραση. Οι μάχημες μονάδες είναι θαυμάσιο εργαλείο για να ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ κρατών πελών, ώστε να υπάρχουν περισσότερα κίνητρα για την ανάπτυξη ικανοτήτων και για την κατάρτιση και εκπαίδευση και για την τυποποίηση μεταξύ αυτών των ομάδων που συμβάλλουν σε μια επιχείρηση πώς μπορεί μία μάχημη μονάδα να χρησιμοποιηθεί. Ως μία πρώτη δύναμη και πρόσφατα, πριν από δύο μήνες, η ομάδα χωρών της Βαϊμάρης υπογράμμισε σε ένα έγγραφο τη σημασία που έχει η πιθανή χρήση μιας μάχης μονάδας για την έναρξη της επιχείρησης και για μεγαλύτερη τυποποίηση των μέσων συμπεριλαμβάνωμένη της ευθυγράμμιση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τυποποίηση, την πιστοποίηση και την εκπαίδευση. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ε, ένα μέσο ad hoc σε περίπτωση που μια επιχείρηση επιδεινώνεται όπου μια αποστολή ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη και θα χρειάζεται να αποχωρήσουν οι δυνάμεις σε, μια, σε ένα πεδίο επιχειρήσεων. Επίσης, προσωρινά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως γέφυρα που θα συνδεθεί με την αρχική έναρξη της επιχείρησης και όπως γνωρίζετε ποτέ δεν χρησιμοποιήσαμε αυτές τις μάχημες μονάδες, αλλά μπορεί να αποτελέσουν γέφυρα και πρόσφατα έγινε αυτό ε, στην Κεντρική Αφρική έκαναν τη γέφυρα μεταξύ ε, της, ε, των Αφρικανικών δυνάμεων και την ανάπτυξη και την αναβάθμιση ε, των δυνάμεων του ΟΗΕ. Επίσης, από καιρούς καιρών υπάρχει μια αμφιλεγόμενη συζήτηση σχετικά με την πιθανή χρήση των μονάδων αυτών ως εφεδρικών δυνάμεων στα πλαίσια των ήδη προσχεδιασμένων ή εξελισσόμενων στρατητικών επιχειρήσεων. Το παράδειγμα της Βοσνίας Αζεγοβίνης, όπου προκύπτει μάλιστα από κύριους καιρών αυτή η συζήτηση, αλλά δεν έχει καταλήξει και δεν αποτελεί μέρος της έννοιας των μαχήμων μονάδων. Ποιοι είναι οι περιορισμοί της χρήσης μιας μάχημης μονάδας. Κυρίως από στρατιωτική άποψη και από τη σκοπιά των, της διαχείρισης των προσδοκιών. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτές οι μονάδες έχουν περιορισμένη εμβέλεια. Εξορισμού δεν μπορεί να είναι γενικός μηχανισμός που να καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αλλά μπορεί ε, να χρησιμοποιείται, να είναι πολύ χρήσιμος μηχανισμός. Οι περισσότερες μάχημες μονάδες μας που βρίσκονται στο Μητρό δεν είναι κοινέ. Λοιπόν, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και ε, θέλουμε να υπόψη και τα εναέρια και θαλάσσια μέσα ε, είναι περιορισμένη χρήση τους από χρονικής απόψεως. Λοιπόν, στις περισσότερες περιπτώσεις, από στρατηγική και στρατηγική πλευρά, πρέπει να σκεφτόμαστε ποια θα είναι η συνέχεια και θα πρέπει να προβλέψουμε και τη συνέχεια μαζί με την εκκίνηση, μαζί με την δραστηριοποίηση των μάχημων μονάδων. Στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται σύντομη προσαρμογή των μάχημων μονάδων στην, σε, μια, ε, σε ένα πεδίο επιχειρήσεων, αν είναι θερμές ή όχι περιοχές, ανάλογα θα γίνει και η προσαρμογή. Κυρίως για το πρώτο θέμα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του 2013 ανέθεσε ε, στην Υπηρεσία Εξωτερική Δράσης και εν μέρη ε, στο στρατιωτικό επιτελείο να προωθήσουν αυτά τα όρια. Και αναπτύξαμε αυτή την έννοια και αρχίσαμε να καλούμε τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν σε αυτό το τομέα. Τι σημαίνει να σπρώξουμε τα όρια. Εισαγάγαμε μία επιπλέον κατηγορία ετοιμότητας που είναι χαμηλότερη από εκείνη των μαχήμων μονάδων, αλλά υψηλότερη από εκείνη τη κανονική διαδικασία δημιουργίας των δυνάμεων. Και αυτό έγινε αποδεκτό από τα κράτη-μέλη. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να έχουμε επιπλέον εναέριες δυνάμεις, θαλάσσιες και χερσαίες δυνάμεις που να περιληφθούν σε αυτόν τον κατάλογο και τα κράτη-μέλη δημιουργούν αυτά τα μητρώα. Το τελικό προϊόν θα πρέπει να είναι μια πιο ευέλικτη χρήση των μαχήμων μονάδων, ώστε να μπορούμε να, τα προσαρμο... να τις προσαρμόζουμε καλύτερα σε μια δεδομένη στρατηγική κατάσταση είτε είναι πιο συγκεκριμένη, είτε ευρύτερη και συνεπώς αυτά τα στοιχεία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε από τις επιπλέον μάχημες μονάδες. Επίσης, α, α, βελτιώσαμε την ετοιμότητα και την έγκαιρη προειδοποίηση με, την, ε, με το Horizon Screening. Στην πράξη, ήδη σε τακτική βάση, ξεκινώντας με, με την εφηβετική περίοδο, καλούμε τους διοικητές αυτών των μονάδων να μας κάνουν την εκτίμησή τους σχετικά με την επιχειρησιακή κατάσταση της Ευρώπης και βεβαίω συμπεριλαμβανομένων των εστιών όπου έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις. Ε, κάνουμε πολλάξ πολιτικές ασκήσεις που οργανώνονται από τις χώρες πλαίσιο. Η πρώτη πολλάξ διεξήχθη πριν από 1,5 χρόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο ε, που ήταν η χώρα πλαίσιο. Η Σουηδία επίσης έκανε μια πολύ καλή πόλαξε και αυτή θα γίνει κοινή πρακτική προκειμένου να ενισχυθεί το συνέστημα ότι πρέπει να λαμβάνονται αποφάσεις έγκαιρα σε πολιτικό επίπεδο και να βελτιώνεται η έγκαιρη προειδοποίηση. Τώρα η χρηματοδότηση. Στα πλαίσια του προγράμματος ε, Αθηνά παρατείναμε τις ισχύουσες ρυθμίσεις για άλλα δύο χρόνια, οι οποίες τι είναι. Οι στρατηγικές ε, εναέριες μεταφορές, αεροπορικές μεταφορές θα γίνονται κατά 60% από τις ε, ε, κυβερνητικές δυνατότητες και 40% από άλλες. Επίσης, θέλω να αναφέρω τη σημασία της συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ για τα θέματα αυτά. Θέλουμε περισσότερες κοινέ προδιαγραφές και εργαζόμαστε για να τις έχουμε. Θα βοηθούσαν πολύ να έχουμε κοινή πιστοποίηση και να έχουμε κοινή εκπαίδευση και ασκήσεις. Με το συγκρότημα μάχης του Βίζεγκραντ που είναι σε φάση σύστασης θα το επιδιώξουμε. Υπάρχουν εναλλακτικέ λύσεις για να, σε αυτά τα συγκροτήματα μάχης για τις ε, περιπτώσεις που σας περιέγραψα. Για μια γενιά μάλλον όχι, με μια εξαίρεση. Αν υπάρχει ένα μεγάλο κράτος αναφοράς, κράτος πλαίσιο που πολύ σύντομα να μας ε, υποβάλει ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Θα μπορούσε να συμβεί. Δεν έχει συμβεί ποτέ για επιχειρήσεις της Ένωσης, αλλά δεν το αποκλείω. Δεν υπάρχει ε, όμως καμία δυνατότητα εάν τα κράτη-μέλη δεν μας δώσουν επιπλέον δυνάμεις. Αυτό μπορεί να γίνει με βάση το άρθρο 44 της συνθήκης που είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή. Δεν έχω σαφή μηνύματα για το τι θα μπορούσαν να δεχτούμε με βάση το άρθρο 44 τα κράτη-μέλη ως μέσο για ταχεία αντίδραση. Κατά λίγο. Μεταξύ τρία σημεία. Πρώτον, η ταχεία αντίδραση είναι περίπλοκο καθήκον και πολύ ευρύτερο από απλώς η χρήση συγκροτημάτων μάχης. Δεύτερον, τα συγκροτήματα μάχης είναι στα πλαίσια αυτά πολύ σημαντικό εργαλείο. Αλλά ένα συγκρότημα μάχης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλες τις αποστολές, όλα τα καθήκοντα. Και τρίτον, η λήψη πολιτικών αποφάσεων και η δημοσιοποίησή τους πρέπει να είναι στο επίπεδο της βούλησης των κρατών μελών να μας δώσουν τις αναγκαίες δυνατότητες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ στρατηγέ. Δεν έχουμε το συντονιστή του ΕΛΚΕ. Κατάλαβα ότι ο κύριος Τέτινα θα τον εκπροσωπήσει. Έχετε τον λόγο. Είμαι από την Πράγα. Άρα είμαστε γείτονες. Πριν από πολύ καιρό, πολλά χρόνια, είχα έναν ε, ξάδελφο που είχε το ίδιο επώνυμο με εσάς, Βόστολσομπια. Είναι λοιπόν ε, διαδεδομένο τσεχικό επώνυμο. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν ότι είμαστε μακρινοί συγγενείς. Αλλά δεν είναι ο μόνος λόγος για τον οποίο νομίζω ότι μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε στον άλλον. Ερώτηση λοιπόν. Συζητούσαν προηγουμένως και εδώ και μήνες το θέμα της Ουκρανίας και ο κύριος Ποροσέγκο, πρόεδρος της χώρας, πρόσφατα είπε ότι θα καλωσόριζε κάποια μορφή συνεργασίας ε, του Ουκρανικού στρατού με τις ευρωπαϊκές ε, ενοπλές δυνάμεις. Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοούσε αλλά η ερώτησή μου είναι εάν υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις ε, στην Ευρώπη που θα μπορούσαν να κάνουν κοινέ ασκήσεις με τις Ουκρανικές ενόπλες δυνάμεις Ξέρω ότι προετοιμάζεται στρατιωτικές ασκήσεις ως ΝΑΤΟ με τον Ουκρανικό στρατό. Υπάρχουν ε, σκέψεις ε, ευρωπαϊκές πολιτικές δυνάμεις, ε, στρατιωτικές δυνάμεις να διεξάγουν τέτοιες κοινέ ασκήσεις. Ευχαριστώ, λέει ο κύριος ε, Πάσκου, για την παρουσίασή σας στρατηγιά. Θέλω διευκρινίσει για τα εξής. Όταν έχετε μία μονάδα που πρέπει να εισέλθει σε ένα χώρο επιχειρήσεων, τότε πρέπει να προετοιμάσετε άλλες τρεις για να μπορεί να γίνει εναλλαγή. Αυτό ισχύει και τα συγκροτήματα μάχης. Είπατε ότι πρέπει να σκεφτείτε μετά την πρώτη είσοδο τι θα γίνει μετά. Γιατί αυτό δημιουργεί και μια σειρά πολιτικά προβλήματα. Δεύτερον, Είπατε ότι τα συγκροτήματα μάχης δεν ε, μπορεί να είναι ενός μεγέθους για όλες τις καταστάσεις. Γιατί οι καταστάσεις μπορεί να είναι περίπλοκες. Αλλά προβλέπετε το ενδεχόμενο καταστάσεων να αποφασίσουμε να εισαχθεί ένα συγκρότημα μάχης και μετά όταν πρέπει να το αντικαταστήσουμε ή να το συμπληρώσουμε, να έχουμε προβλήματα, γιατί μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι κλιμάκος, υπάρχουν πολιτικές αντίρρησεις. Οπότε τι κατάσταση θα προκύψει. Τι θα θυσιάσουμε τις δυνάμεις που έχουν ήδη εισαχθεί. Αναφερθήκατε στις πόλεξ, τις πολιτικές ασκήσεις. Δεν το ήξερα. Υποθέτω ότι γίνονται σε επίπεδο κράτους, όχι σε επίπεδο συμβουλίου. Αλλά καταλαβαίνω την προστιθέμενη αξία του συντονισμού και νομίζω και ότι τα κοινοβούλια των συμμετεχόντων κρατών θα έπρεπε να συνεννοούνται. Γιατί όλοι θα έπρεπε να εγκρίνουν, όλα αυτά τα κοινοβούλια θα έπρεπε να συμφωνήσουν για την εισαγωγή δυνάμεων. Δύο άλλα. Α, όχι, μια άλλη ερώτηση. Έχουμε χώρες στο βορρά της Ευρώπης, είπατε ότι έχουν ε, ειδικέ ε, ρυθμίσεις ε, όπου έχουν και αεροπορικές δυνάμεις που συμμετέχουν ενώ αλλού δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Για τις βόρειες χώρες Επειδή λοιπόν είναι σε καλύτερο επίπεδο προπαρασκευής ε, σκέφτεστε να χρησιμοποιήσετε αυτές τις δυνάμεις κατά προτεραιότητα γιατί αυτό θα διευκόλυνε. Αυτοί δηλαδή θα ήταν ε, μονάδες από το βορρά, θα ήταν οι πρώτες που θα εισήγοντο σε μια επιχείρηση. Και μετά να έρθουν οι δυνάμεις από νότιες χώρες. Θα μπορούσε να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Και τέλος. Είπατε ότι μπορεί να υπάρξει ένα σημαντικό κράτος πλαίσιο, κράτος αναφοράς, που θα ήταν διαδεθειμένοι να εισέλθουν πρώτοι. Αλλά νομίζω ότι αν ε, υπάρχει ένα τέτοιο κράτος, ε, πιστεύω ότι θα προτιμούσε να παρέμβει μόνο του και όχι σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Άρα πρέπει να βρούμε άλλες λύσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πάσκο. Κύριος Φανόρντεν. Ευχαριστώ στρατηγέ. Ευχαριστώ και σας καλωσορίζω. Είστε εξαιρετικός, ε, αξιωματικός και σίγουρα οποιοδήποτε καθήκον ε, θα το φέρετε εις πέρας πολύ καλά. Αλλά δυστυχώς νομίζω ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα στρατιωτικά καθήκοντα δεν εξυπηρετούν τίποτα και είναι ε, σπατάλη πόρων. Αυτό, αυτή η έννοια του συγκροτήματος μάχης Μα δεν είναι ενωσιακή πρωτοβουλία, δεν είναι ενωσιακή έννοια. Είναι βρετανική έννοια. Ήταν ε, ένας τακτικός σχηματισμός μάχης που αρχίσαμε να χρησιμοποιούμε στη δεκαετία του 70. Θα θυμάστε τον αρχικό και ανέφικτο στόχο να έχουμε 60.000 άνδρες που να μπορούν να αναπτυχθούν ανα πάσα στιγμή. Αλλά το συγκρότημα μάχης, η έννοια εισήχθη στην Ένωση ως ένα υποκατάστατο για να ρίξουμε στάχτη στα μάτια. Ποτέ δεν έχει χρησιμοποιηθεί. Δεύτερον, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει συμπληρωματικές στρατιωτικέ δυνατότητε. Όταν διαβάζει κανεί για αυτά τα συγκροτήματα μάχη, νομίζει ότι είναι επιπλέον δυνάμει. Μα όχι βέβαια. Είναι απλέ δυνάμει που ήδη υπάρχουν στου εθνικού μα στρατού. Αυτές οι δυνάμεις μπορούν να φέρουν εις πέρας εθνικές ή νατοικές αποστολές. Όπου προκύψει κρίση, φυσικά δεν χρησιμοποιούνται ενωσιακά συγκροτήματα μάχης. Η πραγματική ταχεία αντίδραση σε κρίσεις προκύπτει πρώτα απ' όλα από τα έθνη που έχουν δυνατότητα να το κάνουν και δεύτερον από ε, συνασπισμούς των βουλωμένων, αυτών που επιθυμούν δηλαδή να συμμετάσχουν, και τρίτον από το ΝΑΤΟ που έχει μία δύναμη 5.000 με αεροπορική κάλυψη, με ειδικέ δυνάμεις, με στοιχεία εχμής που είναι σε θέση να αναπτυχθούν σε 48 ώρες μετά τη λήψη της πολιτικής απόφασης. Θα πρότεινα ότι το συγκρότημα μάχης είναι ένα όνομα για να ισχυριστούμε ότι έχουμε κάποια στρατιωτική δυνατότητα ως Ένωση στην πραγματικότητα. Εάν δεν υπήρχε η ενωσιακή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, κανείς δεν θα το είχε προσέξει. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Εκτός, εκτός, ότι θα βοηθούσε αντί να αποπροσανατολίζονται από αυτή την πολιτική θα μπορούσαν να επικεντρώσουν περισσότερο τις δυνάμεις του στο ΝΑΤΟ. Έχουμε 22 κράτη-μέλη της Ένωσης που είναι επίσης κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και η Αυστρία και η Φιλανδία και η Σουηδία μπορούν να συμμετάσχουν, όπως συχνά κάνουν, σε νατοικές στρατιωτικές ασκήσεις και να συμμετάσχετε πλήρως. Αυτή είναι η συνεργασία που απαιτείται. Δεν χρειαζόμαστε άλλου είδους μηχανισμούς, δομές για να έχουμε συνεργασία Ένωσης και ΝΑΤΟ. Και τέλος, εάν θέλει να βοηθήσει η Ένωση, ίσως, ίσως, θα μπορούσε να έχει ένα συμπληρωματικό ρόλο, δηλαδή μη στρατιωτικέ δυνατότητες. Αλλά δεν θα πρέπει να παίζει σε αυτό το στρατιωτικό παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριο Σαμπάιος. Η κυρία Σαμπάιος. Είμαι Σουηδή. Και συμμετείχα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όταν λαμβάνονται αποφάσεις ε, για τα συγκροτήματα μάχης. Έχουν ε, δοθεί πάρα πολλά χρήματα για τα συγκροτήματα μάχης και χαίρομαι ιδιαίτερα που τα χρήματα αυτά δεν πήγαν χαμένα. Τα συγκροτήματα μάχης είναι ιδιαίτερα δαπανηρά, αν μου επιτρέψετε να πω, και αποτελούν ένα θέμα συζήτησης πολιτικής στις χώρες Βέλη. Το αν θα πρέπει δηλαδή να υπάρχουν τέτοια συγκροτήματα μάχης ή όχι λαμβάνοντας υπόψη τα κονδύλια που απαιτούνται. Η συζήτηση αυτή συνεχίζεται πάντως στη χώρα μου. Θα ήθελα να σας κάνω μερικές συγκεκριμένες ερωτήσεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στο έγγραφο που κυκλοφόρησε και που αναφέρει ότι υπάρχουν πέντε διαφορετικές, διαφορετικά σενάρια ή εκδοχές. Μιλήσατε για πέντε σενάρια τα οποία απαιτούν μια στρατηγική παρέμβαση. Η αντίδραση. Ένα από αυτά αφορούν την επίλυση συγκρούσεων, αλλά δεν έχει εξηγηθεί επαρκώς. Θα ήθελα να μου πείτε σε τι πλαίσιο αναφέρεστε, πότε θεωρείτε μία, ότι μία στρατιωτική αντίδραση απαιτείται. Ύστερα, τι θα πρέπει να γίνει πριν αυτή την επέμβαση, πριν από τη φάση της επίλυσης, της σύγκρουσης θα πρέπει να υπάρχει και μια στρατηγική εξόδου από αυτή την σύγκρουση έτσι ώστε να μην αφήσουμε μια χαοτική κατάσταση στα σημεία που έχει γίνει η παρέμβαση. Στο έγγραφο αυτό παρέχεται και μια εξήγηση σχετικά με το θέμα της διαδικασίας της ταχείας αντίδρασης και το πώς είναι οργανωμένη. Από ό,τι καταλαβαίνω, μέρος της πολιτικής αξιολόγησης δεν θα αφορά πλέον τη διαδικασία όταν μιλάμε για θέμα διαχείρισης κρίσεων. Θα επιθυμούσα να μου πείτε τι ακριβώς εννοείτε. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρχει μία στρατιωτική αντίδραση αν δεν υπάρχει και μία στρατιωτική στρατηγική. Πώς θα πάμε, πώς θα το κάνουμε, πώς θα αποχωρήσουμε. Αναρωτιέμαι επίσης ως προς το θέμα της, ε, των αποφάσεων που λαμβάνονται από τα εθνικά κοινοβούλια. Γιατί τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να παίζουν ρόλο στην διαδικασία αυτή λήψης αποφάσεων για την αποστολή δυνάμεων. Είναι μια παρατεταμένη, σημαντική διαδικασία, γιατί αυτοί που λαμβάνουν τις αποφάσεις, τα κοινοβούλια δηλαδή, είναι υπεύθυνα για τα όσα συμβαίνουν. Είτε είναι για καλό είτε για κακό. Οι πολιτικοί είναι εκείνοι που φέρουν το βάρος της ευθύνης σε τελική ανάλυση. Είναι λοιπόν σημαντικό η διαδικασία να είναι η ε, ενδεδειγμένη. Αναρωτιέμαι αν τα προβλήματα θα μπορούσαν να επιληθούν με ένα σωστό κείμενο ή αν θα συνεχίσουν να εμένουν. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την πολιτική διαδικασία η οποία συνεπάγεται κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Μπάνκρα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου είναι... Ε, μπορείτε να μου εξηγήσετε πώς είναι προγραμματισμένη αυτή η στρατηγική airlift, στρατηγικό airlift. Εδώ εμπλέκονται 16 ε, ε, χώρες. Ε, εδώ στο 2006 θα μπορούσε να θεωρηθεί λογικό, αλλά λαμβάνοντα υπόψη τα όσα συνέβησαν σήμερα, ας σκεφτούμε την περιοχή της Μαύρης Θάλασσας. Εγώ είμαι Ευρωπαίος πολίτης, αλλά ε, μεταράζω τα όσα άκουσα για την Ατλαντική Συμμαχία και τα συγκροτήματα μάχης, καθώς και για την παροχή αεροσκαφών για στρατιωτικούς σκοπούς. Η ασφάλειά μας, ε, συνεπώς, εξαρτάται από μία ρωσική εταιρεία αεροσκαφών. Πώς θα μπορούσατε να το εξηγήσετε αυτό, τι σχέση έχει με τη σημερινή κατάσταση και πώς αξιολογείτε τη στρατηγική της Ρωσίας και των σχέσεων με την ε, Ατλαντική Συμμαχία και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. υποθετικά πώς θα μπορούσατε να περιγράψετε τις δυνητικές περιοχές όπου θα έπρεπε να χρησιμοποιηθούν άμεσα ομάδες ταχείας αντίδρασης δηλαδή να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες λήψης αποφάσεων ή συνεργασίας Θα πρέπει παράλληλα να οριστεί και το τελικό αποτέλεσμα. Υποθετικά μιλώντας, πού νομίζετε ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μία ισορροπία και να επιτευχθεί μία ομόφωνη αντίδραση. Και με την Ατλαντική Συμμαχία έχουμε προβλήματα όπως υπόθηκε. καταβάλλονται προσπάθειες και μέσα στην Ατλαντική Συμμαχία σε μια προσπάθεια συσχετισμού. Πώς η συνεργασία, πώς θα ορίζατε λοιπόν την πραγματική δυνατότητα δράσης. Thank you very much. Thank you for... Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ για την ευγενική εισαγωγή που κάνατε. Μου θυμίζει το πόσο όμορφη πόλη είναι η Πράγα, γιατί έχω και εγώ συγγενείς εκεί. Τώρα, στις ερωτήσεις σας. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχει πολιτική απόφαση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση για να προωθεί μια στρατιωτική διάσταση στην αντιμετώπιση της κρίσης της Ουκρανίας. Παρόλα αυτά, υπάρχουν διμερώς χώρες μέλη που υποστηρίζουν σε διαφορετικό βαθμό την Ουκρανία για την εξαγωγή ασκήσεων. Θα ήθελα να προσθέσω ότι συνεχίζεται η συνεργασία μας με την Ουκρανία. Αυτό έχει σχέση με την ε, ΠΑ και όπως γνωρίζετε η Ουκρανία ήταν και ε, ε, συνέβαλε και συμβάλλει στην κοινή πολιτική άμυνας. Αυτό αποτελεί μια βάση για συνεργασία. Βεβαίως έχουμε πλήρη συνείδηση και καταλανοούμε ότι αυτή τη στιγμή η Ουκρανία βρίσκεται αντιμέτωπη με άλλα σοβαρά προβλήματα που ξεπερνούν τα πλαίσια της κοινής πολιτικής ε, ασφάλειας. Υπάρχουν ε, οι απαιτήσει της Ουκρανίας για αυξημένη συνεργασία. Αυτά, ε, αυτά τα αιτήματα εξετάζονται σε ενωσιακό πλαίσιο. Θα μπορούσε θεωρητικά, δεν έχει λυθεί κάποια απόφαση, να δοθεί κάποια στήριξη στην αποστολή που ήδη ε, έχει σταλεί στην Ουκρανία. Κύριε Πάσκουνα, έρθω τώρα στα δικά σας ερωτήματα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την εκπεριτροπή σε δράση των συγκροτημάτων μάχης, δεν έχει προγραμματιστεί αυτή η εκπεριτροπή δράση των ε, συγκροτημάτων. Βεβαίως, θα πρέπει να προγραμματίσουμε για μία μεγαλύτερη περίοδο δράσης των συγκροτημάτων. Δεν υπάρχει στρατηγική αποχώρηση μετά από δύο, μετά από τέσσερις μήνες. Από την αρχή όμως θα πρέπει να πούμε ότι το θέμα δεν αφορά μόνο τα συγκροτήματα μάχης, μόνο τις στρατιωτικές δυνάμεις. Αφορά τα μέσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μια στρατηγική εξόδου και να την προσδιορίσουν. Βεβαίως, Εάν επιθυμείτε, για να αναφερθώ σε αυτό που είπατε, το να διατηρηθούν οι δυνάμεις σε μια περιοχή, θα πρέπει να γίνει κάτι. Εάν χρησιμοποιηθεί ένα συγκρότημα μάχης, θα αλλάξει ο αριθμός, θα αλλάξει ο όγκος μετά από τέσσερις μήνες. Ενδεχομένως θα υπάρξει και μια ανάγκη ενδυνάμωσής του και αυτό βεβαίως θα έχει επίπτωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό το θέμα. Τώρα, το θέμα της κλιμάκωσης. Δεν θα έλεγα ότι η απόφαση χρήση ή μη χρήση ενός συγκροτήματο μάχη παρεμποδίστηκε με το σκεπτικό ότι θα μπορούσε να υπάρξει αύξηση της κλιμάκωσης στα πλαίσια τη ΠΑ. Ξεκίνησε από μία αξιολόγηση κινδύνων πολιτικών μεταξύ των άλλων. Παρεμποδίστηκε και από ένα άλλο σκεπτικό. Ξεκινήσει το 2008. Από μια ε, παρέμβαση σε επίπεδο ταξιαρχίας από στρατιωτική άποψη όμως θα μπορούσε να είναι, ε, να είναι η αρχική δύναμη και μετά να ακολουθήσει η ταξιαρχία. Δεν ετέθη λοιπόν θέμα ταξιαρχίας ε, ή περισσότερων δυνάμεων. Δεν ήταν αυτό που μας οδήγησε στην απόφαση ε, να καταφύγουμε στα συγκροτήματα μάχης. Η πολιτική άσκηση βεβαίως έχετε δίκιο, ε, αποτελείται από χώρες μέλη, αλλά όλο και περισσότερο συμμετέχουμε σε αυτό για να μπορέσουμε να ε, δώσουμε σε συμβουλές μας, να παρουσιάσουμε την άποψή μας σε διάφορες περιπτώσεις. Αυτό θα ενδυναμωθεί και οι χώρες μέλη καταφέρνουν να έχουν ένα εθνικό ακροατήριο από όλες τις χώρες μέλη που συμμετέχουν. Το θέμα που θέσατε για τις βόρειες χώρες και τη Μεσόγειο, τις μεσογειακές χώρες, ε, νομίζω ότι πάει πολύ πιο κάτω από την στρατιωτική επιφάνεια. Έχει σχέση με την προσαρμογή ενός συγκροτήματος μάχης. Αυτό θα μπορούσε να προκύψει με διαφορετικούς τρόπους. Ακούσαμε στις αρχές της χρονιάς ε, ότι ε, αφορά τα θέματα άμυνας. Να τίθεται το ερώτημα τι νόημα θα είχε να επαναπροσανατολιστεί η σύνθεση των συγκροτημάτων μάχης το, εκείνο που πυροδότησε όμως αυτή τη συζήτηση ήταν τα κοινά συμφέροντα. Βεβαίως υπάρχει και ένα σημαντικός πολιτικός κίνδυνος το να δημιουργηθούν ρογμές ε, μέσα στην κοινή πολιτική. Αυτό βεβαίως το θέμα ε, έχει μπει λίγο στο παρασκήνιο. Θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ με την παρατήρησή σας ε, ότι μεγάλες χώρες ε, θα δράσουν μόνες τους. Υπάρχει μια σχέση, μια διασύνδεση με το άρθρο 44 και αυτό οδηγεί σε μια σύγχυση σχετικά με το 44. Υπάρχει η αίσθηση ότι αυτό θα μπορούσε, ότι θα ε, πρέπει να γίνει εκ των υστέρων μια πολιτική επιβεβαίωση. Γι' αυτό το λόγο είναι υποσυζήτηση ακόμα το θέμα. Ο κύριος Φανόρντεν έφυγε, αλλά χαίρομαι για τη διευκρίνηση των συγκροτημάτων μάχης. Πρόκειται για μία έννοια στρατιωτική και όχι πολιτική. Είναι ο όρος στρατιωτικός. Τώρα, να σας πω ότι η κοινή πολιτική άμυνας επιλαμβάνεται νέων περιοχών, νέων θεμάτων. Αυτό δεν αφορά τα συγκροτήματα μάχης. Υπάρχουν αποστολές ε, κατα, ε, ε, εξάσκησης και ενημέρωσης. Το κόστος, ναι, ναι, έχετε δίκιο. Θα έπρεπε ο μηχανισμός Αθηνά να αναθεωρηθεί Σε ό,τι αφορά τα πέντε σενάρια, υπάρχει και ένα σενάριο πρόληψης συγκρούσεων. Μπορώ να πω ότι το συγκρότημα μάχης έχει κάποιο ρόλο να διαδραματίσει. Ένα τέτοιο σενάριο όμως θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε κάτι όπου θα απαιτείται μία ταχεία αντίδραση από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανεξάρτητα από το τι θα κάνουμε σε στρατιωτικό πλαίσιο συνδέεται άμεσα με ευρύτερες πολιτικές σκέψεις. Και στις συζητήσεις που γίνονται εν ώψη του Συμβουλίου της Δευτέρας, το PFC, είτε το πολιτικό πλαίσιο για την ολοκληρωμένη προσέγγιση, αποτελεί μία εύγλωτη απόδειξη του τι προσπαθούμε να κάνουμε. Και αυτό καθορίζει το ρόλο των στρατιωτικών μέσων και όχι το αντίθετο. Εγώ θα πήγαινα ακόμα πιο πέρα και θα έλεγα ότι υπάρχει μία ισχυρή όση για τη χρήση στα συγκροτήματα, των συγκροτημάτων μάχης, κάτι που είναι κατανοητό, αλλά η επιθυμία του προσφυγής στα συγκροτήματα μάχης δεν θα πρέπει να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα. Θα πρέπει να ενταχθεί σε ένα πλαίσιο και μπορεί να γίνει. Για παράδειγμα, η στρατηγική παρουσία σε μία περιοχή δεν θα πρέπει να προσδιορίζεται από το μέγεθος του συγκροτήματος μάχης. Ενδεχομένως χρειάζεται και κάτι περισσότερο. Αυτό είναι απάντηση στην ερώτησή σας σχετικά με τη στρατηγική αποχώρησης. Αυτή βεβαίως θα μπορούσε να παραδοθεί η σκητάλη σε άλλες δυνάμεις, αλλά αυτό εντάσσεται σε μια ευρύτερη διαδικασία. Ας πούμε, είναι υπάρχει η διαδικασία στην ε, Κεντρική Αφρική με, τις Ηνωμένες, με Ηνωμένα Έθνη, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκινάει να διαδραματίζει έναν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Καταφέραμε να κάνουμε, ρίξουμε αυτές τις γέφυρες και τώρα περνάμε σε έναν μη εκτελεστικό ρόλο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα επιτυχού στρατηγικής αποχώρησης ή εξόδου. Εδώ υπάρχουν και, έμειναν εκτός στοιχεία που αφορούν ε, τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, έτσι ώστε πάρθηκαν ταχύτερα οι αποφάσεις. Βεβαίως δεν, μπορούν, δεν, μπορούν, δεν μπορεί να εξαλειφθεί, να μην υπολογιστεί η ε, διαδικασία αυτή, αλλά σε ό,τι αφορά την πολιτική πλευρά, προσθέσαμε στοιχεία έτσι ώστε να γίνει πιο ολοκληρωμένη η εικόνα. ενώ αμβλύνουμε τις διαδικασίες στρατηγικών επιλογών. Αυτό παραμένει αναγκαίο, αλλά θα μπορούσε να ενσωματωθεί πολύ πιο γρήγορα και καλύτερα. Αν υπάρχει ανάγκη θα πρέπει να ε, αντιμετωπιστεί με ένα διαφορετικό τρόπο, να υπάρχει ε, να συνυπολογιστεί το θέμα της διαχείρισης κρίσεων. Ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα από στρατιωτική άποψη Τα έλεγα ότι υπάρχει κάποια δυσκολία. Το θέμα δεν αφορά μόνο έναν κατάλογο, είναι ότι τα χρειαστούν χρόνια ολόκληρα το ενδιάμεσο αυτό διάστημα. Και πάλι θα πρέπει να ρωτήσουμε τις χώρες μέλη εάν είναι διατεθειμένες να συμβάλλουν σε επίπεδο συγκροτημάτων μάχης. Η πραγματική πρόκληση εδώ είναι ότι η διαδικασία αυτή η έπρεπε να κινηθεί μεταξύ της υιοθέτηση μιας άποψης και της εφαρμογής. Δηλαδή μπορεί να δοθεί η άδεια ε, έναρξης μιας διαδικασίας εάν υπάρχουν οι απαραίτητα, απαραίτητα συγκροτήματα. Ξέρω από τις περισσότερες χώρες μέλη ότι είναι εφικτό να υπάρξουν τέτοιες ταχείες διαδικασίες, παρόλα αυτά παραμένουν ε, μία πρόκληση. Στην ερώτησή σας, εάν έχουν σχέση τα κοινοβούλια, ναι, ε, έχουν. Τώρα αναφεθήκατε ε, ε, σε μια προσωρινή λύση. Υπάρχουν συμβάσεις. Είναι μια εμπορική λύση. Αυτή τη στιγμή ε, έχουν γίνει σεβαστές αυτές, οι, έχουν προσυπογραφεί αυτές οι συμβάσεις. Εμείς εξαρτώμεθα από αυτό το είδος του αεροσκάφους. Γιατί δεν, έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά ε, ε, ε, πολλά αεροσκάφη όπως έχουν τα Αντόνοφ. Υπάρχουν Αυτά είναι θέματα που αφορούν και το επιτελείο στο Eindhoven. Υπάρχουν και άλλα θέματα συντονισμού. Αυτό βεβαίως ξεπερνάει τα πλαίσια του άλλη. Επανεξετάζουμε ορισμένα θέματα και εξετάζουμε άλλες δυνατότητες. Τώρα, δυνητικές, ε, ε, δυνητικό πλαίσιο που θα μπορούσαν ε, να συμβούν ορισμένα πράγματα. Κέντρο Αφρικανική Δημοκρατία, εκεί υπάρχει το σωστό μέγεθος. Υπήρξε και μία πολύ γοργή ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων. Αποφασίσαμε να μην χρησιμοποιήσουμε τα συγκροτήματα μάχης. Δίχως να επισέλθουμε σε λεπτομέρειες, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα χρήσης ε, των συγκροτημάτων μάχης στο μέλλον όχι ως μοναδική λύση, ως αρχική λύση για να επανέλθω στο ερώτημα που πετετέθη από τη Σουηδία. Ένα θέμα που εξετάζουμε με τους υπεύθυνους των συγκροτημάτων μάχης αφορά την παρέμβαση σε μια κατάσταση όπου μία αποστολή βρίσκεται αντιμέτωπη με μία κλιμάκωση ή με μία δύσκολη κατάσταση εκεί θα μπορούσε να ε, δώσει κάποια στήριξη το συγκρότημα μάχης. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα που ετέθη πριν από λίγο σχετικά με το Σάλις και τα Αντώνο. Δίχως άλλο, υπάρχουν τα κατάλληλα αεροσκάφη τα οποία παράγονται στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Είδα φωτογραφίες ε, αεροσκαφών Αντόνοβ με, με την Ουκρανική σημαία ή το χαρακτηριστικό σήμα. Δεν ξέρω αν υπάρχει περίπτωση να επανεξεταστούν οι συμβάσεις ή αν θα μπορούσαμε να εξετάσουμε τις υπάρχουσες δυνατότητες. Γιατί αυτό το σημαίνει ότι θα πρέπει να δείξουμε ότι υποστηρίζουμε αυτή την άποψη. Ήταν ιδέουσα και ίσως όμως τώρα θα πρέπει να επανεξετάσουμε τις αποφάσεις μας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Αυτά είναι εθνικά ουκρανικά αεροπλάνα. Αυτές οι συμβάσεις υπογράφηκαν από τα κράτη-μέλη. Δεν υπάρχει ρόλος των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, ε, αυτό θα πρέπει να το σκεφτούν τα κράτη-μέλη, αφορούν τα κράτη-μέλη. Για πολλά κράτη-μέλη δεν θα είναι εύκολο να επαναχωρήσουν από τα όσα έχουν κάνει. Διότι όπως είπα υπάρχει έλλειψη στρατηγικού airlift παγκοσμίω. Και μάλιστα αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες προτεραιότητες ανάπτυξης δυνατοτήτων που έχουμε. Και ελπίζω και ότι τα κράτη-μέλη της Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν αυτό το θέμα και αυτές τις ελλείψεις. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Εάν όχι, ευχαριστούμε πάρα πολύ στρατηγέ, ειλικρινά, για την παρουσία σας εδώ. Ενημερώνω τα μέλη και τους καλεσμένους μας ότι πριν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Ιουνίου έχουμε την πρόθεση να συζητήσουμε στην ημερησία διάταξη σε πολλά θέματα ε, της Επιτροπής μας, τις ικανότητες, τις στρατιωτικές ικανότητες και της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας και κατόπιν θα γίνει η ενημέρωση των Υπουργών Άμυνας, διότι ο ρόλος τους σε αυτό το τομέα είναι πολύ σημαντικός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ όλα τα μέλη. Σας υπενθυμίζω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα τη Δευτέρα στις 20 Απριλίου το απόγευμα. Είσαστε πρόσδεκτοι. Λύνεται η συνεδρίαση.